Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι. Αρχίζουμε. Θα ήθελα να καλωσορίσω τους ε, καλεσμένους της κυρίας Μίλλερ, που είναι μέλη της Βαβαρικής Ένωσης Γεωργών. Καλώς ήρθατε. Περνάμε στις ψηφοφορίες. Ελπίζω να έχετε φέρει μαζί στις ηλεκτρονικές κάρτες. Το πρώτο θέμα αφορά την έγκριση του σχεδίου σύστασης ε, για τη δεύτερη ανάγνωση ε, για τον κανονισμό Συμβουλίου και Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου προκειμένου να απαγορευτούν μερικές δράσεις που αφορούν την υγεία των ζώων στη κτηνοτροφία. Κύριε Σελιμόβιτς, θέλετε το λόγο. Παρακαλώ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Χαίρομαι ιδιαίτερος που καταλήγουμε εδώ μετά από τόσο χρονοβόρα διαδικασία. Και θα προτιμούσα να μην κάνω κανένα σχόλιο, ελπίζοντας ότι θα υπερψηφίσουμε την ε, σύσταση αυτή, γιατί είναι το επιστέγασμα μιας δεκαετούς ε, προσπάθειας ε, εργόδους. Και θα ήθελα να ευχαριστήσω θερμά την προκάτοχο και να εκφράσω την ελπίδα ότι θα διεκπαιρώσουμε εσύ σήμερα το έργο της. και δεν υπάρχουν πια προβλήματα. Ελπίζω απλώς ότι θα υπερψηφίσουμε το σχέδιο σύστασης. Δεν έχουν κατατεθεί τροπολογίες, οπότε θα ψηφίσουμε με ονομαστική κλίση. Ψηφίσουμε το σχέδιο σύστασης. Άρχεται η ψηφοφορία. Ψηφίσατε όλοι. Τέλος ψηφοφορίας. Πρώτη είναι, γι' αυτό την κράτησα ανοιχτή λίγο παραπάνω. Εγκρίνεται. Καταπληκτικό το αποτέλεσμα. Πανψηφί εγκρίνεται το σχέδιο σύστασης. Σημειώνουμε, λέει ο πρόεδρος, ε, το σχόλιο σα, αλλά δυστυχώ δεν το ακούσαμε γιατί ήταν εκτό μικροφώνου. Όπως σας είπα και χθε η ψηφοφορία της Έκθεση Αγγιλέρα αναβλήθηκε για τη 15η Μαρτίου και σας εξήγησα χθε για ποιο λόγο. Περνάμε στο σημείο 8, την πολιτική συνοχή στις ορεινές περιοχές Ευρωπαϊκή Ένωση. Ο συντάκτης γνωμοδότηση είναι ο κύριος Μισελ Νταντά, γιατί η αρμόδια επί τη ουσία επιτροπή είναι η Επιτροπή Περιφερειακής Ανάπτυξης. Νομίζω ότι ο κατάλληλο να μα κάνει την εισαγωγή είναι ο εισηγητής μας, ο κύριος Νταντά. Θέλετε το λόγο? Δεν χρειάζεται καν. Πολύ ωραία, οπότε μπορούμε να περάσουμε στην ψηφοφορία επί των τροπολογιών. Ξεκινάμε με τη συμβαστική τροπολογία 6. τις αρχές της κοινή γεωρικής πολιτικής ε, για τις ορεινές περιοχές. Θα ψηφίσουμε ηλεκτρονικά τη συμβαστική τροπολογία υπαριθμών 6. Άρχεται η ψηφοφορία. Τέλος ψηφοφορίας. Περνάμε τώρα στη συμβαστική τροπολογία 3. Άρχεται η ψηφοφορία, ηλεκτρονικά και πάλι, συμβαστική τροπολογία 3. Τέλος ψηφοφορίας. Εγκρίνεται και μπορούμε να περάσουμε στη συμβαστική τροπολογία 4. για το συντονισμό των κοινοτικών δράσεων και ταμείων. Άρχεται η ψηφοφορία ηλεκτρονικά και πάλι παρακαλώ. Τέλο ψηφοφορίας. Ψηφίζουμε τώρα την τροπολογία 58. Διανατάσσεως της χειρός. Ποιο είναι υπέρ τη 58. Κατά. Απορρίπτεται. Συμβαστική τροπολογία 9. Απλούστευση της ΚΑΠ και του διοικητικού άχθους. Ηλεκτρονικά ψηφίζουμε. Παρακαλώ, άρχεται η ψηφοφορία. Τέλος ψηφοφορίας. Ευχαριστώ. Εγκρίνεται η συμβαστική 9 και περνάμε στη συμβαστική τροπολογία περιθμών 5 τις μακροπεριφέρειες ε, και τις ε, στρατηγικές για τις ορεινές περιοχές. Άρχεται η ψηφοφορία ηλεκτρονικά, παριθμό 5 συμβαστική τροπολογία. Τέλος ψηφοφορίας. Συμβαστική τροπολογία 15 τώρα. Άρχεται η ψηφοφορία. Αφορά τον τουρισμό και τη φυσική και παραδοσιακή πολιτιστική κληρονομιά. Τέλος ψηφοφορίας. Εγκρίνεται και περνάμε στη συμβαστική τροπολογία 13. Κλίμα και περιβαλλοντικές πτυχές. Άρχεται η ψηφοφορία ηλεκτρονικά για την 13 συμβαστική τροπολογία. Τέλος ψηφοφορίας. Ομόφωνα εγκρίνεται. Και περνάμε στην τροπολογία 67. Διανατάσσει τη χειρό ψηφίζουμε. Ποιο είναι υπέρ τη τροπολογία 67. Κατά. Απορρίπτεται. Και περνάμε στη συμβαστική τροπολογία 7. Α. Αποσύρεται. Την 70 ψηφίζουμε. ποιο είναι υπέρ. Τροπολογία 70, Dortmund και Des. Ποιο είναι κατά. Εγκρίνεται η 70. Τροπολογία 71, Νόικλ. Ποιο είναι υπέρ. Κατά. Απορρίπτεται. 73. Πρώτα όμως θα κάνουμε ηλεκτρονικό έλεγχο για την τροπολογία 71. Άρχεται η ψηφοφορία. Τροπολογία 71, Νόικλ. Τέλος ψηφοφορίας. Ωραία. 73 τώρα, Διανατάσσω της χειρός. Ποιος είναι υπέρ της 73, κατά. Απορρίπτεται. Και περνάμε στη συμβαστική τροπολογία περιθμών 7, που αφορά το δεύτερο πυλώνα. Άρχεται η ψηφοφορία. Τέλος. εγκρίνεται. Συμβαστική τροπολογία 8, υποπρόγραμμα για τα όρη. Άρχεται η ψηφοφορία της συμβαστικής τροπολογίας 8. Τέλος ψηφοφορίας. Εγκρίνεται και ψηφ... περνάμε στη συμβαστική τροπολογία 9 ε, ναι, λέει ο 10 ε, συγγνώμη. Υλικέ και ψηφιακές υποδομές και δημόσιες υπηρεσίες. Άρχεται η ψηφοφορία. Εγκρίνεται η συμβαστική 10. Και περνάμε στη συμβαστική τροπολογία 11. Επιμόρφωση και κατάρτιση. Άρχεται η ψηφοφορία ηλεκτρονικά για την 11. Τέλος ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. Περνάμε στην τροπολογία 106. Διανατάσεις της χειρός ψηφίζουμε. Ποιος είναι υπέρ της 106. Ωραία κατά. Απορρίπτεται. Τροπολογία 101. Ποιος είναι υπέρ. Κατά. Απορρίπτεται. 111. Ποιος είναι υπέρ. Κατά. Απορρίπτεται. Περνάμε στη συμβαστική τροπολογία 17. Ψηφίζουμε ηλεκτρονικά. Αφορά την παραγωγή γάλακτος στις ορεινές περιοχές. Άρχεται η ψηφοφορία. Τέλος ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. εγκρίθηκε η 17, πολύ σημαντική για την παραγωγή γάλακτος. Πέραμε στη συμβαστική τροπολογία 16, δασοκομεία. Άρχεται η ψηφοφορία της, τροπολογίας, της συμβαστικής τροπολογίας 16. Τέλος ψηφοφορίας της 16. Εγκρίνεται και αυτή. Συμβαστική τροπολογία 12 τώρα, που έχει τίτλο «Ρόλος των γυναικών». Άρχεται η ψηφοφορία για την συμβαστική 12. Τέλος ψηφοφορίας. Εγκρίνεται 114 Διανατάσσω της χειρός. Ποιος είναι υπέρ της τροπολογίας 114. Ευχαριστώ κατά. Απορρίπτεται. 118. Ποιος είναι υπέρ. Κατά. Απορρίπτεται. Συμβαστική τροπολογία 14. Τοπικές αγορές και βραχία αλυσίδα ανεφοδιασμού. Ε, σήματα ποιότητας. Άρχεται η ψηφοφορία. Τέλος της ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. Τροπολογία 135 τώρα. Ποιο είναι υπέρ διανατάσσεως της χειρός. Πρόκειται για την τροπολογία Ντεκάστρο. ποιο είναι υπέρ. Εγκρίνεται 135. 136 τώρα, Χόιμπουχ. Ποιο είναι υπέρ. Κατά. Απορρίπτεται. 137. ποιο είναι υπέρ. Κατά. Ηλεκτρονικός έλεγχος για την 137 της ψηφοφορία. Τέλος ψηφοφορίας. 19 υπέρ 23 κατά απορρίπτεται. 129. Ποιος είναι υπέρ της τροπολογίας 129. Κατά. Απορρίπτεται. Τροπολογία 143. Ποιος είναι υπέρ. Κατά. Απορρίπτεται. Τροπολογία 140. Ποιος είναι υπέρ. Κατά. Απορρίπτεται. Περνάμε στις ε, αιτιολογικές σκέψεις και λοιπές παραγράφους καθώς και στο προήμιο. Τροπολογία 1 για την αιτιολογική σκέψη α του κ. Νταντά. Ποιο είναι υπέρ, εγκρίνεται. Τροπολογία 2. Υπέρ. Εγκρίνεται. Τροπολογία 3. Υπέρ. Εγκρίνεται. 4. Υπέρ. Εγκρίνεται. Τροπολογία 5. Υπέρ. Εγκρίνεται. Τροπολογία 6. Υπέρ. Εγκρίνεται. 7. Υπέρ. Εγκρίνεται και αυτή. Περνάμε στη συμβαστική τροπολογία 1. Οι στόχοι της Ευρωπαϊκής Ένωσης ε, σε ό,τι αφορά τη γεωργία στις ορεινές περιοχές. Άρχεται η ψηφοφορία. Τέλος. Εγκρίνεται. Συμβαστική τροπολογία 2. Προκλήσεις στις ορεινές περιοχές. Άρχεται η ψηφοφορία. Τέλος ψηφοφορίας. Άρχεται η ψηφοφορία, λέει ο πρόεδρος πάλι. Τέλος ψηφοφορίας. Πρόκειται για τη συμβαστική τροπολογία 2. Λυπάμαι αμφιλιαρό. Τέλος ψηφοφορίας. Ψηφίσουμε το σύνολο της γνωμοδότησης ε, μετά τις, τις τροπολογίες. Ψηφίζουμε ηλεκτρονικά την τροποποιηθήσα γνωμοδότηση. Άρχεται η ψηφοφορία. Τέλος ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. Σας ευχαριστώ όλους και κυρίως το συντάκτη γνωμοδότησης, τον κύριο Νταντάν. Θέλετε κύριε Νταντάν μήπως το λόγο τώρα. Μάλιστα. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Θα ήθελα να ευχαριστήσω αρχικά τους ασκιώδεις και τους βοηθούς τους, ε, με τους οποίους νομίζω ότι είχαμε μια πολύ καλή συνεργασία. Επιτρέψτε μου να ευχαριστήσω και την ομάδα της ε, γραμματείας ε, της Κοινοβουλευτικής μας Επιτροπής και σας ευχαριστώ όλους για τα αποτελέσματα της ψηφοφορίας. Συμφωνούμε και υπερθεματίζουμε τις ευχαριστίες σας κύριε Νταντά. Πολύ σημαντική η γνωμοδότηση, γιατί συνεχώς μιλούμε για την ανάγκη στήριξης ε, των ορεινών περιοχών, προκειμένου να μπορέσουν να αναπτυχθούν οικονομικά, να συνεχίσουν την ε, παραγωγή γάλακτος, να, ε, να στηριχθούν και οι γυναίκες, ο ρόλος των γυναικών. Το Μάρτιο θα ψηφίσει η Αρμόδια Επιτροπή Ρέγγι και θα περάσει το θέμα στην Ολομέλεια του Απριλίου. Πέραμε τώρα στο σημείο 9. Ανταλλαγή απόψεων με εκπρόσωπο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής από τη Γενική Διεύθυνση Γεωργίας για την ευθυγράμμιση και την απλούστευση του δευτερογενούς νομοθεσίες στον τομέα των απορροκυπευτικών και του ίνου. Εκπρόσωπος Ευρωπαϊκής Επιτροπής είναι ο κύριος Γιώστ Κόρτε, τον οποίο καλωσορίζουμε μαζί με το επιτελείο του. Και θα του δώσω το λόγο για να μας παρουσιάσει τα βασικά στοιχεία, τις βασικές πτυχές ε, του κατεξουδότηση κανονισμού για τα απορροκυπευτικά. Πολύ σημαντικό θέμα που έχει ζωηρό ενδιαφέρον. Επίσης το θέμα του κατεξοδότηση κανονισμού για, την, για τις προδιαγραφές ε, της θέσης εμπορία και της επισήμασης του ίνου και τα δύο θέματα είναι πολύ σημαντικά και περιμένουμε τις απόψεις Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Στόχος είναι η ενοποίηση και η απλούστευση του νομοθετικού πλαισίου για τους δύο αυτούς τομείς των απορροκυπευτικών και του ίνου. Βρίσκονται και οι δύο κανονισμοί σε προπαρασκευαστικό στάδιο. Παρόλο, το Παρόλο που το θέμα των κατεξοδότηση πράξεων έχει προχωρήσει πολύ περισσότερο. Από τη στιγμή που θα εγκριθούν, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θα σκίσει το δικαίωμα που έχει να εκφέρει αντιρρήσεις κατά το κατεξοδότηση πράξεων για τα προκυπευτικά μέσα σε δύο μήνες. Ε, σε ό,τι αφορά την εκτελεστική πράξη για τον Ίνο, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο δεν έχει δικαίωμα άρνηση Αυτά επί της διαδικασίας, επί της ουσίας θα μας μιλήσει ο εκπρόσωπος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, ο κύριος Κόρτε. Παρακαλώ κύριε Κόρτε, έχετε το λόγο. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε αξιότιμα μέλη. Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω για την πρόσκλησή σας να παρευρεθώ στη σημερινή σας συνεδρίαση για να σας ομιλήσω για ορισμένα σημαντικά κατά τη γνώμη μας ζητήματα τα οποία εξετάζει αυτή την περίοδο η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και πιο συγκεκριμένα θα ήθελα να αναφερθώ ε, στο παράγωγο δίκαιο, κατεξοδότηση και εφαρμοστικές πράξεις που εκπονούμε για τα εθνικά προγράμματα στήριξης για τον Ίνο και τα απορροκυπευτικά δύο επιμέρους ζητήματα όπου έχουμε προχωρήσει αρκετά στις εργασίες μας. Και μετά, Πρόεδρε, επιτρέψτε μου επί τη ευκαιρία να διευκρινίσω και τι συνεχιζόμενες εργασίε, εκεί που δηλαδή που δεν έχουμε προχωρήσει αρκετά, σε ό,τι αφορά τα πρότυπα θέσεις εμπορία και ε, επισήμανσης. Ε, εν γέννη, Όντως και στο Κοινοβούλιο έχουμε δει πολλές κοινοβουλευτικές ερωτήσεις, επιστολές, ε, σημαντικό ενδιαφέρον υπάρχει και από το Συμβούλιο αλλά και από τα ενδιαφέρουνα μέρη, ιδίω από τον ε, παραγωγικό κλάδο. Θα ήθελα λοιπόν να διευκρινίσω που βρισκόμαστε και σε αυτό το τρίτο σημείο, όπου ακόμα δεν υπάρχει κείμενο το οποίο εκπονείται. Και πριν αρχίσω να σας μιλώ για τα προγράμματα στήριξης ε, του Ίνου, να σας πω και δύο λόγια για το σκοπό μας. Γιατί δηλαδή κάνουμε ό,τι κάνουμε. Είναι σημαντικό να κατανοήσουν και τα μέλη το υπόβαθρο. Αυτή τη στιγμή υπό την βασική πράξη ε, για την κοινή οργάνωση αγοράς, κανονισμός 1308 του 2013, Βεβαίως, ε, στο πλαίσιο της τελευταίας ε, μεταρρύθμισης ε, της κοινή γεωργικής πολιτικής, είχαμε περίπου 200, 200 κανονισμούς παράγου δικαίου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Στην πλειονότητά του ακόμα είναι εκτελεστικέ πράξει. Όμω, δυνάμει τη συνθήκη Λισαβόνα και τη ίδια της βασική πράξη, ο 1308 θα πρέπει να λισαβονοποιηθεί, αυτή η τρομερή λέξη βεβαίω. Πρέπει δηλαδή να κάνουμε τη διάκριση μεταξύ καταξιδότηση και ε, εκτελεστικών πράξεων από την άλλη. Αυτό είναι ο κινητήριο μοχλός όλων των εργασιών μας. Βεβαίω, εφόσον πολλοί από αυτού τους κανονισμού είναι αρκετά παλαιοί, προσπαθούμε, σε συνεργασία και με εσά και με τα κράτη-μέλη, να αξιοποιήσουμε αυτή την ευκαιρία. Ε, να τα απλουστεύσουμε, να τα εξυγχρονίσουμε, ε, να βρούμε μια λογική συνεκτική προσέγγιση σε όλους τους κλάδους. Και αυτό είναι κάτι το οποίο είναι ιδιαίτερα σημαντικό για ε, τον Επιτροπό μας. Όμως το υπόβαθρο, ο πυρήνας αυτής της διαδικασίας είναι η συμμόρφωση και εναρμόνιση με τη συνθήκη της Λισαβόνας. Και εσείς τα ξέρετε όλα αυτά σε ό,τι φοράει και τον οργανισμό για την κοινή οργάνωση της αγοράς. Ο σκοπός ε, που έχει θέσει ο ίδιος ο Επίτροπος για την διαδικασία απλούστευσης παύλα λησοβονοποίησης είναι να πέσουμε από του 200 κανονισμούς περίπου σε 40. 40 κατά εξουδότηση και εκταλιστικές πράξεις στο σύνολό τους. Και αυτό από πλευρά Ευρωπαϊκής Επιτροπής είναι πολύ λογικό. Εντάσσεται και στο πλαίσιο της Επιτροπής Juncker και των στόχων της για την καλύτερη ρύθμιση και νομοθεσία και μεγαλύτερη επικουρικότητα. Δεν σημαίνει απορρίθμιση. Δεν θα ήθελα που δεν είναι να χρησιμοποιήσω αυτόν τον όρο. Αλλά θα επανέλθω. Για να πάει καλά αυτή η διαδικασία, ήδη από το 2014 έχουμε ξεκινήσει μια καινοτόμη διαδικασία με ευρύτατη συμμετοχή. Καλούμε πολλούς ε, ενδιαφερόμενους από την αρχή για να μας μιλήσουν ε, για τις απόψεις τους Ξέρω ότι δεν είναι δικές μου υποθέσεις, Πρόεδρε, αλλά πρέπει παρόλα αυτά να αναφέρω ότι είμαστε λίγο απογοητευμένοι στη Γενική Διεύθυνση Γεωργίας για το γεγονός ότι η συμμετοχή του Κοινοβουλίου σε διαδικασία δεν είναι πολύ καλά οργανωμένη μέχρι τώρα. Πάντα καλούμε τους εμπειρογνώμονές σας μαζί με τους εμπειρογνώμονες των κρατών μελών σε αυτές τις συναντήσεις, όμως η συμμετοχή είναι αρκετά χαμηλή. Δεν ξέρω βεβαίως αν ε, έχω το δικαίωμα να σας ε, το επισημάνω, αλλά θα ήθελα να εξετάσουμε που κατά πόσο μπορούμε να εμπλέξουμε τα μέλη του Κοινοβουλίου ε, στα αρχικά στάδια της διαδικασίας. Δεν έχει τόσο νόημα τώρα που έρχομαι εγώ εκ των υστέρων σχεδόν να σας παρουσιάσω τα, παρουσιάσω έχουν συμβεί τον τελευταίο χρόνο. Αυτά ήθελα να πω εν είδη εισαγωγής. Κάθε 6-7 μήνες, νομίζω, σας στέλνουμε έναν κατάλογο των κατεξουδότηση πράξεων που προετοιμάζονται για να γνωρίζετε ότι τα εξετάζουμε και αυτό και πάλι αποτελεί πρόσκληση προς εσάς για να συμμετάσχετε στη διαδικασία. Ξέρετε ότι τελικά γίνεται υιοθέτηση των κατεξοδότηση πράξεων από την Κομισιόν, όμως μετά υπάρχουμε μία δίμηνη περίοδο ε, κοινοβουλευτικού ελέγχου και είναι κρίσιμη σημασία η δική σας συμμετοχή και εμπλοκή. Τώρα για να περάσω στο πρώτο από τα ζητήματα που έχετε θέσει. Τα εθνικά προγράμματα στήριξη στον ε, τομέα του ίνου. Είναι πολύ σημαντικά ε, προγράμματα και από πλευρά πολιτικού υποβάθρου. Ιδιαίτερα επιτυχή, για ζωή σας στοιχεία, από το 2009 τα προγράμματα στήριξη του ίνου με χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης είχαν πολύ μεγάλο αντίκτυπο στις εξαγωγέ ίνου εκτός Ένωσης. Το 2015 έχουμε σημειώσει αύξηση 9% στην αξία των εξαγωγών και 3% σε απόψη όγκου. Είναι λοιπόν πολύ σημαντικό για το εμπορικό συζύγιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Κατά μέσο όρο από αυτά τα προγράμματα διατίθεται ποσό περίπου 1,1 δις ευρώ κάθε χρόνο. Πολύ σημαντικά λοιπόν αυτά τα προγράμματα, γι' αυτό θα πρέπει και η οργάνωση και η νομοθεσία ε, που τα διέπει να είναι πολύ καλά οργανωμένη. Τώρα εξετάζουμε και εκτελεστική και καταξιδότηση πράξη για αυτό το ζήτημα. Ε, προϊόν και όρια δύο ετών εργασιών με τους εμπειρογνώμονους που ανέφερα και ελπίζουμε να ψηφιστεί στην Επιτροπή ε, πολύ σύντομα η, η εκτελεστική πράξη, και η καταξιδότηση πράξη μέσα σε ορισμένε εβδομάδες και μετά βέβαια θα υποβληθεί σε εσά και στο Συμβούλιο για ε, την ε, εξέταση. Τώρα, για τα βασικά ζητήματα αυτών των δύο πράξεων, Προσπαθήσαμε πάνω απ' όλα να εισαγάγουμε σαφήνεια σε ό,τι αφορά ε, τον αποχαρακτηρισμό ε, του πρώτου πυλώνα, των προγραμμάτων δηλαδή στήριξη στον πρώτο πυλώνα και των προγραμμάτων που υπάρχουν στο δεύτερο πυλώνα για τον Ίνο. Βεβαίω υπήρξε και έκθεση του ελεγκτικού συνεδρίου με πολλές επικρίσεις και αξιοποιήσαμε την ευκαιρία για να αποφύγουμε οποιοδήποτε είδους διπλή χρηματοδότηση, όπου ο εμπορευόμενος ε, θα επωφελείται και του πρώτου και του δεύτερου προγράμματος στήριξης ε, από τον πρώτο και τον δεύτερο πυλώνα, το οποίο δεν επιτρέπεται από τον νόμο. Έχουμε προσπαθήσει να ξεχρονίσουμε και σε ό,τι αφορά τις ε, προκαταβολές, τις αποζημιώσεις δαπανών και ολόκληρο το σύστημα ελέγχων και κοινοποιήσεων. Τώρα, για να περάσω στο δεύτερο ε, σημείο, τα απορρικεπτικά. Και εδώ έχουμε καταξιδιώτηση πράξη και εκτελεστική πράξη. Περίπου 10 συναντήσεις είχαμε με εμπειρογνώμενες ε, των κρατών μελών από το 2014 και μετά μέχρι και σήμερα. Και είχαμε και πολλές επαφές με, τους, ε, με τα διάφορα μέρη στην Κόπα Κοζέγκα και εκπροσώπους του κλάδου όπου όπως ξέρετε οργανώνεται σε οργανώσεις παραγωγών και διακλαδικές. Ελπίζουμε να υιοθετηθεί η καταξιότητα της πράξης μέσα σε, στους επόμενους μήνες. Εξαιρετικά σημαντικό στοιχείο για τα προγράμματα στήριξης που έχουμε σε αυτόν τον πυλώνα και τα οπορικευευτικά είναι ακριβώς οι οργανώσεις παραγωγών. Μάλιστα όλη η στήριξη για αυτόν τον κλάδο διοχετεύεται μέσω αυτών των οργανώσεων και έτσι αυτή η καταξιότηση πράξη είναι ιδιαίτερα λεπτομερής, γεμάτη λεπτομερέστα τους κανόνες για το πώς αυτές οι οργανώσεις παραγωγών θα πρέπει ε, να δομούνται και πώς μπορούμε εμείς να τις χρηματοδοτήσουμε με έναν τρόπο που να συνάδει και με τις ε, νομικές μας ε, διατάξεις. Και αυτό είναι εξαιρετικά σημαντικό και πάλι, γιατί έχουμε έρθει ε, αντιμέτωποι και με οικονομικές διορθέωσεις στο παρελθόν σε πέντε κράτη-μέλη, ακριβώς εξαιτία ε, αυτών των οργανώσεων παραγωγών και όλα αυτά πρόσφατα. Υπάρχει λοιπόν ζήτημα σε αυτό το σημείο και προσπαθούμε να το διευκρινίσουμε με αυτούς τους κανόνες για να αποφεύγουμε ε, αυτές τις λυπηρές οικονομικές διορθώσεις. Να αναφέρω ορισμένα στοιχεία που έχουμε συμπεριλάβει στο σχέδιο κειμένου. Ελάχιστος αριθμός μελών των οργανώσεων παραγωγών. Αυτή είναι μια σημαντική διάταξη, ε, προκειμένου να αναγνωρίζονται. Και ένα σημαντικό σημείο το οποίο θα επανέλθει και στη συνέχεια νομίζω, η θέση εμπορία των ε, εμπορευμάτων από μέλη εκτός των οργανώσεων παραγωγών. Και υπάρχει και η δημοκρατική λογοδοσία ε, των οργανώσεων παραγωγών και η εξωτερική ανάθεση των δραστηριοτήτων τους. Πολλά από αυτά τα ζητήματα είναι σημαντικά, γιατί αν επιτρέψουμε υπό το ευρωπαϊκό δίκαιο στους παραγωγούς ε, να αποφασίζουν από κοινού για τιμέ, για την πώληση, για την διαχείριση ε, της προσφοράς, προφανώς και υπάρχει έλεγχος από τις αρχές ανταγωνισμού τον, του κράτους μέλους και από τη δική μου Γενική Διεύθυνση Ανταγωνισμού. Πρέπει λοιπόν να διασφαλίσουμε ότι αυτές οι δραστηριότητες βεβαίως και δίνεται δυνατότητα να συμβούν και αυτό προκύπτει από το πλαίσιο μας, το οποίο είναι ιδιαίτερα εύρωστο σε ό,τι αφορά την παρέκκληση από ε, τους κανόνες ανταγωνισμού, μόνο όμως αν τηρούνται αυτοί οι κανόνες και από τα μέλη των οργανώσεων παραγωγών. Και έτσι με αυτού του κανονισμού προσπαθούμε να δώσουμε ώστε το γίνεται μεγαλύτερη σαφήνεια για το τι μπορούν και τι δεν μπορούν να κάνουν. Γι' αυτό, για παράδειγμα, είναι εξαιρετικά ε, δύσκολο να είναι κανεί μέλο οργάνωση παραγωγών και ταυτόχρονα μεμονωμένα να ε, πουλάει κανεί τα προϊόντα του. Δεν γίνονται και τα δύο είτε συλλογικά μέσω τη οργάνωση παραγωγών δραστηριοποιείται κάποιο, είτε είναι πλήρω ε, ιδιωτικό φορέα, αναλαμβάνοντα και τον επιχειρηματικό κίνδυνο. Όμως το να συμμετέχει κανεί και να κάνει και τα δύο κανείς σίγουρα δημιουργεί ένα προβληματισμό. Για να σα δώσω μόνο μία πρώτη γεύση ε, της περιπλοκότητας του ζητήματος, αλλά υπάρχουν και ας πούμε ε, διασυνοριακέ οργανώσεις παραγωγών. Πήγα στη Μαδρίτη πριν μήνε σε μία έκθεση και πραγματικά εντυπωσιάστηκα με το πόσο προηγμένες είναι αυτές οι οργανώσεις και αυτοί οι όμιλοι, γιατί λειτουργούν και διασυνοριακά, όχι μόνο εθνικά και περιφερειακά. Για μα είναι πολύ θετικό που προσπαθούν να οργανώσουν το εμπόριο και με αυτόν τον τρόπο προσπαθούν να του βοηθήσουμε. Μετά, ένα σημείο που επίση είναι πολύ ε, πολύπλοκο και το επεξεργαζόμαστε, περιβαλλοντικέ προδιαγραφέ και όροι που πρέπει να τηρούν οι οργανώσει παραγωγών. Αυτό εντάσσεται και στο διατακτικό του 1308. Υπάρχει λοιπόν ε, όρος ε, για την οργάνωση παραγωγών να εκπονεί και περιβαλλοντικές ε, δραστηριότητες και υπάρχει μια σάφεια για το πόσα μέλη της οργάνωσης παραγωγών θα πρέπει να συμμετέχουν σε αυτές τις δραστηριότητες. Προσπαθούμε να τα διευκρινίσουμε όλα αυτά και να δώσουμε και μεγαλύτερα περιθώρια ευελιξίας στην οργάνωση παραγωγών και να εκπληρώσει αυτούς τους όρους. Τέλος, ένα σημείο το οποίο είναι σημαντικό σε αυτή την νομοθετική πράξη είναι το σύστημα τιμή εισόδου. Στον ίδιο κανονισμό, δεν έχει σχέση με την οργάνωση παραγωγών. Υπάρχουν επίσης λοιπόν διατάξεις στον ίδιο κανονισμό για το πώς θα ελέγχουμε το σεβασμό, του, την τήρηση του καθεστώτος εισαγωγών ε, για τα απορριγευτικά, ιδίω για τι ντομάτε. Έχουμε ένα ε, πολύ πολύπλοκο λοιπόν σύστημα με διάφορες υποχρεώσεις ε, και πιστώσεις ε, απέναντι στο Μαρόκο και προσπαθούμε όλα αυτά να τα απλουστεύσουμε και να ενιοποιήσουμε το ε, σύστημα της τιμής εισόδου. Κάτι το οποίο θα έχετε προσέξει και εσείς είναι ότι θέλουμε να φύγουμε από τον καθορισμό της ε, ημερήσιας ε, τιμής εισαγωγής στην εβδομαδιαία, το SIV στο λεγόμενο. Είναι σημαντικά όλα αυτά για τις ε, τελωνικές μας αρχές και για τους εμπόρους, για να ξέρουν σε ποιο επίπεδο μπορούν να εισέλθουν στην ευρωπαϊκή αγορά χωρίς να πληγούν από έναν απαγορευτικό ε, εισαγωγικό δασμό. Έχουμε κάνει διάφορες ε, προσωμιώσεις, έχουμε μιλήσει και με τους εμπορευομένους και τους ε, ενδιαφερομένους από το Μαρόκο για να φύγουμε από αυτό το σύστημα και να εγκαταλείψουμε το σύστημα ημερήσιου ορισμού του SIV και να περάσουμε σε εβδομαδιαίο ορισμό της τιμής αυτής. Δεν έχουμε λάβει ακόμα απόφαση και τα τρία κύρια κράτη-μέλη ε, που αφορούν αυτό το, το εμπόριο της δομάτας Ισπανία, Γαλλία και Ιταλία και το Μαρόκο, είναι όλοι ικανοποιημένοι με αυτή την πρόταση. Αυτό σημαίνει ότι είτε η Κομισιόν έχει κάνει τεράστιο σφάλμα, είτε ότι μάλλον καλά τα έχουμε πάει και καταφέραμε να βρούμε τη χρυσή τομή. Το εξετάζουμε και μπορούμε να το συζητήσουμε και στο μέλλον. Τέλος, ό,τι αφορά τα ε, πρότυπα θέσεις εμπορία και την επισήμανση, ιδίως ό,τι αφορά τον κλάδο του ίνου. Γιατί εκεί ήταν η πιο έντονο το ενδιαφέρον. Είναι εξαιρετικά σημαντικό να θέσουμε αυτή τη συζήτηση στο κατάλληλο πλαίσιο και πάλι. Σήμερα, υπό τον ίδιο κανονισμό κοινή οργάνωση αγορά, το 1308 του έχουμε υιοθετήσει στο παρελθόν 15 κανονισμούς που θέτουν πρότυπα, θέσεις εμπορία και διατάξεις επισήμανσης. 15 επιμέρους κανονισμούς για πάρα πολλά προϊόντα. Όλοι αυτοί οι κανονισμοί που είναι εκτελεστικές πράξεις θα πρέπει να ευθυγραμμιστούν και να εναρμονιστούν μεταξύ τους. Πρέπει λοιπόν, κανονικά θα είχαμε τουλάχιστον 30 θα πρέπει να του πάσουμε σε εκτελεστική και κατοξιδότηση πράξη. Και έτσι θα είχαμε 30 κανονισμούς. Και πάλι δεν είναι πολύ ελκυστική ιδέα κατά τη γνώμη μα. Έτσι λοιπόν ξεκινήσαμε με κάθε ερεμία να ρωτάμε τους εμπειρογνώμους και τα κράτη-μέλη κατά πόσο θα μπορούσαμε να συγχωνεύσουμε κάποια από αυτά τα κείμενα. Ε, να έχουμε ένα κείμενο που να ισχύει για όλα τα πρότυπα θέσει εμπορία. Να έχουμε τις διατάξεις ε, ελέγχων κοινοποιήσεων όλα τα οριζόντια ζητήματα σε ένα κείμενο και να μην τα επαναλαμβάνουμε ξανά και ξανά. Και βεβαίως προσπαθήσαμε επί τη ευκαιρία να απλουστεύσουμε και να ενιοποιήσουμε κάποιους από αυτούς τους ε, κανόνες. Πρόσφατα μόνο ξεκινήσαμε αυτό το χείρημα, δεν έχουμε προχωρήσει πολύ και δεν υπάρχουν ακόμα συγκεκριμένες προτάσεις, να μην τις περιμένετε σύντομα. Το πιο σημαντικό, σας διαβεβαιώ, ότι ανεξαρτήτως του τελικού αποτελέσματος, αυτές οι διεργασίες δεν ε, αμφισβητούν το πολιτικό συμβιβασμό επί της πολιτικής ε, που αποφασίστηκε και συμφωνήθηκε το 2013 και δεν σημαίνει ότι θέλουμε να τροποποιήσουμε την ουσία των κανόνων της θέσης εμπορία και των σχετικών προτύπων. Δεν υπάρχει καμία πρόθεση λοιπόν να τροποποιήσουμε ε, κάποιες από τις βασικές διατάξεις επισήμανσης του παραγωγικού κλάδου ή άλλα ζητήματα που θα υπονομεύσουν το νομικό πλαίσιο ε, του κλάδου του ίνου. Αυτό το έχουμε ξεκαθαρίσει πολλές φορές κατόπιν ε, οδηγιών που έχουμε λάβει από τον Επίτροπο και το έχουν εφαρμόσει και οι συνάδελφοι. Παρ' όλα αυτά βλέπουμε ότι υπάρχει ανησυχία ε, στον εμπορικό κλάδο, ότι προσπαθούμε να απορριθμίσουμε τον κλάδο ή να εγκαταλείψουμε κάποιους κανόνες. Δεν ισχύει κάτι τέτοιο. Και έτσι αποφασίσαμε υπό το φως όλων των ερωτημάτων που έχουν τεθεί να αξιολογήσουμε και να συνεχίσουμε να αξιολογούμε. Και να εξετάσουμε σε μεγαλύτερο βάθος αυτό το ζήτημα μέχρι να έχουμε όλα τα στοιχεία στη διάθεσή μας για να αποφασίσουμε τι θα πρέπει να γίνει. Τελικά βέβαια. Ίσως θα ήταν εύκολο να μην αγγίξουμε κανένα από αυτούς τους κανόνες. Όταν το συζητούσαμε με τους συναδέλφους μου, για να είμαι στην Επιτροπή πρόσφατα, λέγαμε, μα γιατί να αλλάξουμε κάτι, ας τα αφήσουμε όπως είναι. Όμως, πρέπει, δυστυχώς, <laughs> να το πω έτσι, ε, πρέπει, υπάρχει νομική υποχρέωση να ε, διαχωρίσουμε όλους τους κανονισμούς σε δύο τμήματα. Και κάποια στιγμή ε, ορισμένοι θα διερωτηθούν γιατί έχουμε τόσες εκτελεστικές διατάξεις για όλα αυτά τα στοιχεία. Δεν θα γίνει ε, σύντομα, αλλά κάποιοι θα προσφύγουν στο δικαστήριο και θα πούνε εμένα δεν με δεσμεύει αυτό το στοιχείο, γιατί θα είναι εκτελεστική πράξη, ενώ θα πρέπει να είναι κατεξουσιοδότηση πράξη. Κάποια στιγμή λοιπόν θα πρέπει να υπάρξει αυτός ο διαχωνισμός. Και μια άλλη διαδικασία που θα ήθελα να επισημάνω εδώ. Ορισμένες διατάξεις για τα πρότυπα θέσεις σε εμπορία που αφορούν τον έλεγχο των προτύπων. Σήμερα δεν υπάρχουν συγκεκριμένοι κανόνες στην κοινή γεωργική πολιτική για το πώς θα ελέγχονται αυτά τα πρότυπα. Έτσι, με βάση του κανόνες τη Ευρωπαϊκής Ένωσης, τα κράτη-μέλη είναι αρμόδια για αυτόν τον έλεγχο. Εφόσον δεν ενέχονται πόροι από τον προπολογισμό μας, οι δικές μας ελεγκτικέ αρχές δεν το ιεραρχούν ω προτεραιότητα και δεν υπάρχει και νομική βάση. Τα κρατημέρια λοιπόν πρέπει να προχωρήσουν στου ελέγχου. δεν ξέρουμε πώ ακριβώ γίνεται αυτό και είναι ακόμα ένα λόγος για τον οποίο τρέχει αυτή η διαδικασία στο Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο για τον επίσημο κανονισμό ελέγχων τροφίμων και ζωοτροφών. 882 του 2004. Υπάρχει λοιπόν μια συζήτηση εκεί για το κατά πόσο ο έλεγχος των προτύπων θέσης εμπορία θα συμπεριληφθεί σε αυτόν τον κανονισμό. Νομίζω ότι είναι μια τροπολογία του Κοινοβουλίου. Εάν λοιπόν ε, εγκριθεί αυτή η πράξη και το αναλάβουν οι συνάδελφοι της Γενικής Διεύθυνσης ε, ΣΑΝΚΟ, όχι δική μου, τότε θα έχουμε διαφορετικούς κανόνες για τους ελέγχους. Και αυτό με τη σειρά του ε, θα μας αναγκάσει να εξετάσουμε αυτούς τους 15 κανονισμούς που έχουμε αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει καμία βιασύνη Και πάλι δεν σας λέω ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα υποβάλει προτάσεις σύντομα. Αντιθέτως, όμως, κάποια στιγμή θα πρέπει να καταλήξουμε κάπως αυτή τη διαδικασία. Σας ευχαριστώ πολύ για την προσοχή σας και θα προσπαθήσω να απαντήσω όσο μπορώ πιο πληρέστατα τις ερωτήσεις σας. Σας ευχαριστούμε κύριε Διευθυντά. Θα ακούσουμε τώρα τις παρατηρήσεις και τις ερωτήσεις των ε, Ευρωβουλευτών. Η κυρία Εράνς Γκαρσία. Ευχαριστώ Πρόεδρε και ευχαριστώ την Ευρωπαϊκή Επιτροπή που έχει την καλοσύνη να έρθει και να μας ε, μιλήσει για δύο πολύ σημαντικά θέματα, τα απορροκυπευτικά και τον ίνο. Αλλά με προβλημάτισε πολύ η Ευρωπαϊκή Επιτροπή με την παρουσίαση που έκανε. Στο θέμα των απορροκυπευτικών, θα ξεκινήσω με αυτό. Δεν έγινε λόγος για τις τιμές εισόδου στην αγορά της μαροκινής ντομάτας και των υπόλοιπων προκυπευτικών. Με το προηγούμενο καθεστώς ε, είχαμε διαδοχικές ε, κριτικές επικρίσεις και καταγγελίες από Ευρωπαίους ντοματοπαραγωγούς ε, εξαιτίας των καταχρήσεων που έκανε το Μαρόκο στο προηγούμενο καθεστώς. Γι' αυτό ζητήσαμε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να λύσει αυτό το θέμα που πραγματικά ήταν σκανδαλώδες και κράτησε χρόνια ολόκληρη. Τώρα, για το κρασί θα έπρεπε να έχουμε ένα καλύτερο σύστημα, να αποφεύγουμε τις προηγούμενες καταχρήσεις, αλλά φαίνεται ότι με την έναρξη της μεταρρύθμισης αυτό που συνέβη, ε, το Μαρόκο επινόησε ε, την, ε, την συμπερίληψη και των ντοματών τσέρι στην συνολική εκτίμηση, τον υπολογισμό της τιμής εισόδου της ντομάτας, κάνοντας όμως κατάχρηση, γιατί οι κανονικές ντομάτες φαίνεται ότι έχουν υψηλότερη τιμή από αυτή που πραγματικά έχουν. Δηλαδή έκανε κόλπο το Μαρόκο με το συνυπολογισμό ε, της ε, τσέρι ντομάτας. Αυτό το ζήτησε η τελεί και η Ισπανία να διαχωριστούν οι τσέρι ντομάτες ε, γιατί αυτές έχουν το μεγαλύτερο ανταγωνισμό με τις μαροκινές ντομάτες. Τώρα αν εσείς ε, επιμείνετε στην απλούστευση και στην ευθυγράμμιση αυτό που θα καταφέρετε τελικά είναι να αυξήσετε την ε, πιθανότητα να κάνει κόλπα και καταχρήσει το Μαρόκο. Οπότε διαστρεβλώνονται οι συνθήκες του ανταγωνισμού. Είναι σαν να έχουμε ένα ποδοσφαιρικό αγώνα και στη μία ομάδα να τους ε, κλείνουμε τα μάτια, να τους δέρουμε τα μάτια για να μην μπορούν να βλέπουν πώς διεξάγεται το παιχνίδι. Αυτό φοβάμαι ότι θα είναι το αποτέλεσμα ε, της ε, νέας μεταρρύθμισης. Θα έχουμε συνεχώς καταγγελίες ε, εις βάρος του Μαρόκου για καταχρήσεις του κανονισμού. Και δεν το ζήτησε μόνο η Ισπανία, το ζήτησε και η Ιταλία, το ζήτησε και η Γαλλία. Είναι τρεις οι χώρες μέλη με εντοματοπαραγωγούς που την ίδια περίοδο καταγγέλουν αυτές τις προτάσεις. Επίσης, τι γίνεται με τις αποζημιώσεις για τις αποσύρσεις λόγω της κρίσης στην αγορά. Ούτε καλύπτεται το κόστος παραγωγής καν. Επιτέλους θα πρέπει να γίνει ενημέρωση αυτών των τιμών. Αυτά για τα απορροκυπευτικά. Σε ό,τι αφορά το κρασί, και εκεί ανησυχώ τα μάλα γιατί βλέπω δύο πράγματα εδώ. Στο έγγραφο εργασία ε, εξαφανίστηκαν κάποιοι υπάρχοντες κανόνες. Δεν περιλαμβάνονται στο έγγραφο εργασία ε, πολλοί κανόνες που ισχύουν για τις ονομασίες προέλευσης αυτή τη στιγμή. Τι σημαίνει αυτό, από τη στιγμή που παραλείπονται έχουν καταργηθεί, έχουν εξαφανιστεί. Γιατί έχουν εξαφανιστεί αυτές ε, οι χρήσεις, οι ειδικές χρήσεις για την αγορά προέλευσης ε, ή την χρήση επισήμανσης συγκεκριμένης ε, περιοχής. Γιατί ένα επιτραπέζιο κρασί του Ριβέρα Ντεντουέρο που δεν έχει ονομασία προέλευσης δεν θεωρείται τέτοιο. Ή κάποιο κρασί που δεν παράγεται στη Ριόχα και είναι επιτραπέζιο να αναφέρεται Ριόχα. Νομίζω ότι έτσι παραπλανάται ο καταναλωτής. Δεν νομίζω ότι θέλουμε να τον παραπλανήσουμε. Παρακαλώ. Η αναφορά της γεωγραφικής ένδειξης θα πρέπει να αναφέρεται μόνο στις ονομασίες προέλευσης. Γιατί έφυγε από το κείμενο, παραλήθηκε από το κείμενο το θέμα των παραδοσιακών αναφορών που προηγουμένως συνδέονταν με τις ονομασίες προέλευσης. Θέλετε οι επιτραπέζοι είναι να έχουν τις παραδοσιακές αναφορές για να οδηγούν και να παραπλανούν τον καταναλωτή. Θα σας δώσω ένα τελικό παράδειγμα, το αμπρούσκο. Η ονομασία αμπρούσκο μπορούν να, ε, να περιλαμβάνεται μόνο στα ε, κρασιά ονομασία προέλευσης της Ρωμάνια. Δεν θέλετε οποιοδήποτε επιτραπέζιο κρασί από την Ιταλία να μπορεί να αναφέρει την ονομασία Αμπρούσκο και να νομίζω καταναλωτή ότι πίνει κρασί από την ε, περιοχή Ρωμάνια. Νομίζω ότι παραπλανούμε έτσι τον καταναλωτή και ό,τι παραλήφθηκε από τους προηγούμενους κανόνες θα πρέπει να επαναφερθεί σε αυτό το έγγραφο εργασίας για να μην δημιουργήσουμε την εντύπωση ότι έχουμε απορριθμίσει πλήρως την αγορά. Επίσης, τι δομή αμπελοεινικών κανόνων θα έχουμε. Θα έχουμε ειδικό κανονισμό για τον αμπελοεινικό τομέα σε ένα μόνο έγγραφο ή θα έχουμε κατακαιρματισμό των ε, κανόνων στα διάφορα νομοθετικά κείμενα. Γιατί αν θέλετε σαφή κανονισμό που θα εφαρμόζεται εύκολα και θα ευκολύνει και τους παραγωγούς και τους διανομής ίνου, μάλιστα. Ή μήπως θέλετε να παραπλανήσετε τους πάντες και να δημιουργηθεί ένα συνοθήλευμα κανόνων που κανένας δεν θα καταλαβαίνει τι ισχύει. Ευχαριστώ κύριο Ντόρφμαν. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε και για τη συζήτηση που γίνεται σήμερα το πρωί. Τρία θέματα θέλω να δείξω. Κύριε Πρόεδρε, παρακαλώ να το κοιτάξετε λιγάκι γιατί με εξέπληξε αυτή η εισαγωγική ομιλία του κυρίου Κόρτε. Εδώ και αρκετή ώρα διερωτώ με Πώς είναι δυνατόν όσοι ασχολούνται με τις ε, κατεξουσιοδότηση πράξεις ε, του Κοινοβουλίου να πηγαίνουν στην Κομισιόν και να μην μας ενημερώνουν ποτέ. Ο κύριος Κόρτε λέει ότι ούτε και αυτοί όταν πάνε στην Κομισιόν ενημερώνονται. Άρα αυτό πρέπει να μας προβληματίσει. Κατά τα άλλα, νομίζω ότι οι πρώτες που έκανε ο κύριος Κόρτε σχετικά με την συμμετοχή και την ποιότητα συμμετοχής του Κοινοβουλίου, ότι αυτό πρέπει λιγάκι να μας ε, προβληματίσει και να προβληματιστούμε είναι σωστό να εκπροσωπούμε τα στο επίπεδο που εκπροσωπούμε τα σήμερα. Ο κύριος Κόρτε είπε ότι στις αρχικές φάσεις ε, δεν εκπροσωπεί το Κοινοβούλιο και γι' αυτό συζητιούνται αυτά που συζητιούνται σήμερα εδώ. Αυτά για τον τύπο. Τώρα, για τα, ε, επί της ουσίας, οπωροκυπευτικά, να δείξω ένα θέμα το οποίο ε, αφορά την παραγωγή οπωροκυπευτικών στην Ιταλία. Κοιτάξτε, στην Ιταλία υπάρχει ένα σύστημα όπου ε, μέλη των παραγωγών δεν είναι μεμονωμένη παραγωγή, αλλά συνεταιρισμοί, οι οποίοι συνεταιρισμοί έχουν μικρούς ε, παραγωγούς που είναι μέλη των συνεταιρισμών και σε δεύτερη βαθμίδα αυτοί είναι μέλη των συνεταιρισμών παραγωγής. Στην Ιταλία έτσι είναι οργανωμένο το σύστημα, λειτουργεί πάρα πολύ καλά και νομίζω ότι υπάρχουν πολύ λίγοι τομείς ε, όπου η αγορά των οποροκυπευτικών να είναι τόσο καλά οργανωμένη όσο ε, στην δική μου την περιοχή που πρόκειται για την παραγωγή μήλων. Βλέποντας λοιπόν την πρόταση, με προβληματίζουν ορισμένα πράγματα. Δηλαδή, κατά πόσον ο κανονισμός ε, που ίσχυε μέχρι σήμερα μπορεί να συνεχίσει να ισχύει ως έχει. Διότι το να ανατεθούν κάποιες δραστηριότητες παραγωγής ε, στους ε, συνεταιρισμούς, αυτό αντιμετωπίζεται με τον ίδιο τρόπο όπως η ανάθεση σε τρίτους. Αυτό λοιπόν είναι κάτι τελείως διαφορετικό και μέχρι τώρα αντιμετωπιζόταν και ως ε, κάτι τελείως διαφορετικό. Νομίζω λοιπόν ότι ε, στην περίπτωση αυτή έχουμε ένα πολύ καλά δοκιμασμένο σύστημα που απέδειξε ότι είναι επιτυχές και γι' αυτό λοιπόν πρέπει να το διατηρήσουμε, να εξτάσουμε όλα τα θέματα ε, κάτω από αυτό το πρίσμα να ορίσουμε ακριβώς πότε θα τεθούν όλα αυτά σε ισχύ. Νομίζω και από αυτού αυτή τη στιγμή το σχέδιο δεν είναι ακριβές. Πρέπει να ξεκαθαρίσουμε ότι όλα αυτά θα τεθούν σε ισχύ από την 1η 1 η 17 και το θέμα των ε, μεταβατικών διατάξεων εκκρεμεί. Όσον αφορά τώρα τον ίνο. Κοιτάξτε, το κρασί μπορεί κανείς να το δει είτε μισογεμάτο είτε μισοάδιο. Εγώ πιστεύω η κατεξουσιοδότηση και οι εφαρμοστικές ε, πράξεις ε, προσφέρουν και δυνατότητες απλούστευσης. Αυτή τη στιγμή βιώνουμε την αλλαγή του συστήματος. Σήμερα βιώνουμε όλες τις αλλαγές ε, των διατάξεων παραγωγής για την ονομασία προέλευσης για όλα τα προϊόντα και για το κρασί και αυτά δεν γίνονται πλέον σε εθνικό επίπεδο αλλά στην Κομισιόν. Άρα έχει υπάρξει μια καθυστέρηση που είναι και παράλογη που σημαίνει ότι έχουμε περιπτώσεις όπου πρόκειται για αμελητές αλλαγές των διατάξεων παραγωγής και αυτές εκκρεμούν στην Κομισιόν εδώ και χρόνια γιατί η Κομισιόν δεν έχει τη δυνατότητα να τα ε, επεξεργαστεί αυτά μέσα σε ένα εύλογο χρονικό διάστημα. Νομίζω λοιπόν ότι όλες αυτές οι μικρές, ή αμελητές αλλαγές θα πρέπει να ανατεθούν στα κράτη-μέλη και η Κομισιόν επιλαμβάνεται μόνο των σημαντικών διατάξεων. Δηλαδή νέες διατάξεις για ή νέες διατάξεις για ονομασίες προέλευσης. Με λίγα λόγια, πράγματι, όταν είναι σημαντικές αλλαγές, να γίνονται από την Κομισιόν αν τα εφαρμόσουμε αυτά που σας λέω, θα ελαφρύνουμε την ε, δουλειά της Κομισιόν και θα αναθέσουμε και κάποια, κάποιες αρμόδιες στα κράτη-μέλη που δεν νομίζω ότι υπάρχει πρόβλημα. Όσον αφορά την αναφορά ποικιλιών, συμφωνώ με αυτά που είπε η συνάδελφος Εστεχέρεντ αλλά και ο κύριος Κόρτε δεν τα είπε κατηγορηματικά στην αναφορά του. Όταν πρόκειται για την χρήση ποικιλιών, κυρίως ε, στους επιτραπέζιους ίνους, πριν από κάποια χρόνια είχε υπάρξει κάποιο συμβασμός. Τώρα δεν έχει κανένα νόημα μία κατεξουσιοδότηση πράξη να την ε, επιβάλλουμε και να ξεχάσουμε το συμβασμό που επιτεύχθηκε πολύ δύσκολα στον κανονισμό αγοράς για το κρασί. Δεν πρέπει να αμφισβητήσουμε αυτόν τον κανονισμό, ούτε και θα κερδίσουμε τίποτα αν ένας ε, παραγωγός από την Ισπανία ε, χρησιμοποιήσει την ποικιλία και την ονομασία Λαμπρούσκο τέτοιου είδους ποικιλίε είναι συνδεδεμένες με συγκεκριμένες περιοχές, ε, ισχύουν κυρίως ε, στις ε, καλλιέργειες στο νότο της Ευρώπης, στη Μεσόγειο. Άρα δηλαδή πρέπει να σεβαστούμε το συμβασμό. Αυτές οι ποικιλίε μπορούν να χρησιμοποιούνται και χωρίς αναφορά της ονομασίας προέλευσης. Αυτό να συνεχίσει να υπάρχει. Παρακαλώ λοιπόν η Κομισιόν να το δει λιγάκι το θέμα αυτό και να το συμπεριλάβει στις προτάσεις. Κατά τα άλλα, ε, έχω απόλυτη κατανόηση για το ότι πράγματι πρέπει ε, να υπάρχει ε, περίληψη και συρρήκνωση ορισμένων πραγμάτων, αλλά δεν θέλω αύριο ο παραγωγός να αναγκαστεί στην ετικέτα να γράφει όχι μία ποικιλία αλλά πέντε. Να έχουμε δηλαδή κατά νου την απλούστευση και σε πρακτική εφαρμογή. Ένας οριζόντιος κανονισμός ε, μπορεί να οδηγήσει στο να υπάρχουν πράγματι λιγότερες κατεξιότητες πράξεις, αλλά αν αυτό βοηθάει τελικά τον ε, παραγωγό, ε, αυτό το αμφισβητώ. Κατόπιν τούτου πρέπει να εξετάσουμε και το θέμα της απλούστευσης και κάτω από αυτό το πρίσμα που μόλις τώρα σας παρουσίασα. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πολύ. Είναι πολύ ενδιαφέρουσα και πολύ σημαντική η σημερινή συζήτηση. Ο εκπρόσωπο τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή μα είπε ότι δεν θέλει να μιλήσει για απορρίθμιση. Αν δεν θέλετε να μιλήσουμε για απορρίθμιση, τότε χρειαζόμαστε αποδείξει και στοιχεία ότι αυτή η διαδικασία πλούστευσης με την οποία συμφωνούμε όλοι δεν συνιστά απορρίθμιση. Συμφωνώ με τα όσα είπε η κυρία Ραν όταν αναφέρθηκε στο ζήτημα του ίνου. Γιατί η απλούστευση εδώ έχει λίγο την αίσθηση της απορρίθμισης και θα επηρεάσει και τις επιχειρήσεις και τους καταναλωτές. Σε ό,τι αφορά τα όπορο ο βασικός στόχος πολιτικής είναι η ενίσχυση των οργανώσεων των παραγωγών και κάθε φορά που παίρνω το λόγο σε αυτή την γεωργική επιτροπή λέω ότι ο οργανός παραγωγών είναι το μέσο που θα μας επιτρέψει να επιτύχουμε το σκοπό μας. Και ο σκοπό μας είναι η διασφάλιση ενός αξιοπρεπούς εισοδήματος για τον ε, παραγωγό δεν είναι αυτό ο σκοπό λοιπόν. Όπω ξέρετε, ο τομέας των υπερκευτικών ε, γνωρίζει μεγάλες μεταπτώσεις τιμέ τιμές ε, και αβεβαιότητα. Πρέπει λοιπόν να πάμε πέραν τούτου. Μιλήσατε και για τις τιμές εισόδου. Πρέπει να τι προσαρμόσουμε. Και μιλήσαμε για μια χαρακτηριστική περίπτωση που είναι αυτή τη ντομάτα του Μαρόκου. Δεν ξέρω αν η Ευρωπαϊκή Επιτροπή διάβασε την έκθεση μέλο που εγκρίναμε εδώ για τα απορροκυπευτικά. Πέρασε στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και από την έκθεση είναι σαφέ ότι η κατάσταση στον κράτο αυτό είναι απελπιστική και σε όλη την Νότια Ευρώπη πολλοί καλλιεργητές οπωροκυπευτικών εγκαταλείπουν τις καλλιέργειές τους και εγκαταλείπουν τα κτήματά τους. Η κατάσταση τα απορροκυπευτικά είναι καταστροφική ιδιαίτερα στην Νότια Ευρώπη. Και αν συνεχίσουμε και δεν φροντίσουμε να έχουμε αποδεκτή τιμή για τα προϊόντα τους οι καλλιεργητές, πολύ φοβάμαι ότι μετά από 20 χρόνια, μέσα σε 20 χρόνια θα εξαφανιστεί όλη η παραγωγή απορροκυπευτικών στην Ευρώπη. Οπότε έτσι θα έχουμε γλιτώσει και από το πρόβλημα, αν θέλετε. Αλλά θα συνεχίσουμε την αύξηση των εισαγωγών απορροκυπευτικών από τρίτε χώρε. Και μάλιστα ε, τα προϊόντα αυτά υφίστανται επεξεργασίε με χημικά προϊόντα που εμεί απαγορεύουμε τιμή προεκυπευτικών αυτή τη στιγμή στην Ευρωπαϊκή Ένωση για τους δικού μας παραγωγούς δεν είναι επαρκής για να εξασφαλίσει την παραγωγικότητα και την επιβίωση του κλάδου. Αυτό το λέει η έκθεση μέλου, εδώ έβγαλα από το μυαλό μου. Και υπάρχει και αθέμητος ανταγωνισμός από τρίτες χώρες. Δεν ξέρω αν διαβάσετε την ομολογία του ΔΕΚ ε, από την υπόθεση της Ευρωπαϊκής Ένωσης κατά του Μαρόκου. Γιατί ε, και προϊόντα από τη Δυτική Σαχάρα ε, εξάγει το Μαρόκο. Θα πρέπει να ξέρουμε λοιπόν από πού προέρχονται τα προϊόντα που εισάγουμε και τι ε, συνθήκες ισχύουν εκεί. Επίσης, ε, η τιμή απόσυρσης σε περίπτωση αστάθειας της παραγωγής και οι τιμές που εφαρμόζονται για την απόσυρση ιδιαίτερα σε κρίση όπως με, την, με το εμπάργο της Ρωσίας για προϊόντα όπως ο λωτός ή το ρόδι η τιμή απόσυρσης είναι πραγματικά γελία. Είναι ε, τόσο πενιχρές αυτές οι τιμές που σε καμία περίπτωση δεν εξασφαλίζουν τους γεωργούς. Επίσης, ε, για τις ε, τιμές εμπορίας. Αναφέρεται ότι μια, μια οργάνωση παραγωγών θα γνωρίζει από τη στιγμή της ε, παραγωγής την τιμή της διάθεσης. Μακάρι, αλλά δεν νομίζω ότι ισχύει αυτό, πολλά δε μάλλον που έχουμε και πολλές εισαγωγές. Θα πρέπει να το καλοσκεφτούμε λοιπόν πριν το προτείνουμε. Επίσης, το θέμα των περιβαλλοντικών κριτηρίων. Εγώ ανήκω στους πράσινους στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και εμείς προτείναμε την ανάμειξη των οργανώσεων παραγωγών ώστε να κάνουν επενδύσεις που να βελτιώνουν την περιβαλλοντική πτυχή των, ε, της παραγωγής και των καλλιεργιών τους. Ήδη οι Γεωργοί έχουν κάνει πολλές τέτοιες φιλοπεριβαλλοντικές επενδύσεις ε, και έχουν φτάσει στο οι άνθρωποι. Θα πρέπει, αν θέλουμε να διατηρήσουμε αυτή τη στρατηγική, να προβλέψουμε ενισχύσεις. Και όσοι, γεωργοί ήταν οι καλοί μαθητές και έχουν κάνει τα καθήκοντά τους, να στηριχθούν περαιτέρω για να συνεχίσουν στον καλό αυτό δρόμο. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ κύριε grazie. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε και ευχαριστώ πολύ και τον ε, εκπρόσωπο της Κομισιόν για την παρέμβασή του. Εγώ θέλω να έχω κάποιες διευκρινήσεις, κυρίως όσον αφορά τον ε, τομέα του των απορροκητευτικών και του ίνου. Πρόκειται για τον ε, κανονισμό ο οποίος έχει σχέση με την επισήμανση. Αυτό είναι ένα θέμα που το έφυξαν βέβαια στην συνάδελφοί μου. Σήμερα γνωρίζουμε πολύ καλά, εκόντες άκοντες πρέπει να ασχοληθούμε με αυτό τον κανονισμό διότι έχει αλλάξει η νομική βάση ε, και έχουν προκύψει κάποιες ε, ασάφειες. Νομίζω όμως ότι όσοι ασχολούνται με το κρασί θα πρέπει να καθησυχαστούν ε, πρέπει να τους ζητήσουμε κάποια συγνώμη για το ότι ε, πλέον δεν υπάρχει προστασία για αυτούς. Αυτό ισχύει κυρίως ε, για, τους, για τα προϊόντα με ονομασία προέλευσης. Άρθρο 32. Ερωτώ την Κομισιόν. Πρόκειται για κάποιες ετικέτες κρασιών σε σχέση με την ονομασία προέλευσης. Έγινε λόγος για το κρασί λαμπρούσκο. Ξέρουμε ότι υπάρχουν ε, κάποιες ε, τεχνικές εξελίξεις που καθιστούν απαραίτητο να ανανοηθεί λιγάκι αυτή η ονομασία προέλευσης ε, για να μην υπάρχει κατάχρηση. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή μπορεί να μας εγγυηθεί ότι η κατάσταση όσο έχει σήμερα ε, μπορεί να επιφέρει σε ασφάλεια και να μην υπάρξουν υποχωρήσεις. Δηλαδή, να μην επιτραπεί να συνδέεται ένα προϊόν με την περιφέρεια ή με τις υπόλοιπες ποικιλίε. Αυτό να είναι ένα δικαίωμα το οποίο θα ενισχύεται και επίσης ε, θα υπάρχουν και εγγύησεις για το δικαίωμα αυτό. Ο κύριος Νταντά. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Θα ήθελα πρώτα να ευχαριστήσω τον κύριο Κόρτε, τον εκπρόσωπο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, ε, για τη σαφήνεια με την οποία παρουσίασε τις προτάσεις ε, και την επισήμανση της ανάγκης ε, μεγαλύτερης ανάμειξης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στις εργασίες αυτές. Έχω δύο σχόλια. Καταρχήν, ως προς τον Ίνο, διαπιστώνουμε ότι δεν έχουν προχωρήσει αρκετά οι εργασίε των ίνων σε σχέση με αυτέ για τα απορροκρυφτικά. Εκεί είμαστε πολύ πιο προχωρημένοι. Σε ό,τι αφορά το κείμενο για τον ίνο, σίγουρα θα πρέπει να γίνει κάποια λισαβονοποίηση εντό εισαγωγικών, αλλά θα πρέπει ταυτόχρονα να είμαστε και προσεκτικοί για να μην διακυβεύσουμε τι ε, πολιτικέ συμφωνίε των διαπραγματεύσεων του 2008 και του 2013. Και δεν σας κρύβω ότι μετά τις εξηγήσεις που άκουσα από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, μου ήρθαν στο μυαλό κάποια σχόλια που άκουσα από τους συνοπαραγωγούς στις διαπραγματεύσεις που έγιναν το 2012 και 2013. Έχω την αίσθηση να ακούω εκείνους ε, που ήταν ε, κατά της επανεισαγωγής ε, ενός δικαιώματος παραγωγής. Φυσικά θέλουμε ένα ισορροπημένο κείμενο και όχι μία απλή επανάληψη των προσδοκιών ε, του εμπορικού κλάδου για τον ίνο. Φυσικά ε, χρειάζεται διανομή, αλλά χρειάζεται κυρίως παραγωγή. Και φυσικά ευκρίνεια και σωστή ενημέρωση του καταναλωτή. Για το θέμα των γεωγραφικών ενδείξεων, για παράδειγμα, και της επισήμασης ε, θα πρέπει να βρίσκονται στο ίδιο κείμενο, να αποφευθεί η διασπορά των νομοθετικών διατάξεων σε μια πληθώρα γράφων, κάτι που θα δημιουργήσει το όλο νομοθετικό πλέγμα ακατανόητο για εκείνου που θα χρειαστεί να το εφαρμόσουν. Σε ό,τι αφορά την κοινή οργάνωση αγορά απορριπευτικών, εδώ έχουμε ένα πιο εξεζητημένο κείμενο, σε πιο προηγμένη φάση τη διαπραγμάτευση με το Συμβούλιο. Γνωρίζω τις δυσκολίες που αντιμετωπίζει η Γενική Διεύθυνση Γεωργίας για το θέμα αυτό και θα πρέπει όλοι να βρισκόμαστε σε εγρήγορση και να επαγρυπνούμε ώστε να τηρηθεί το άρθρο 39 της συνθήκης της Λισαβόνας γιατί αυτό επιτρέπει τις εξαιρέσεις ε, από το δίκαιο ανταγωνισμού για τη γεωργία και τη συμπεριλήψη και των οργανώσεων των παραγωγών. Οπότε θα πρέπει η Γενική Διεύθυνση ΚΟΜΠ ε, για τον ανταγωνισμό να αφισβητήσει αυτά που ήδη επιθυμήσαμε και αναδείξαμε στις διαπραγματεύσεις για την κοινή οργάνωση αγοράς στα απορροκυπευτικά. Επίσης θα πρέπει να μεριμνήσουμε ώστε οι νέες απαιτήσεις που θα επιβληθούν στους γεωργούς να μην ε, επιβαρύνουν αντί να απλουστεύσουν όπως δήλωσε ο Επίτροπος ότι είναι το ζητούμενο. Επίσης αναφέρατε μία τριετή διάρκεια. Αυτό δεν συμβαίνει για να γίνεται έλεγχος κάθε χρόνο, αλλά να γίνεται έλεγχος, να γίνεται έλεγχος κάθε τριετία. Αυτό το νόημα έχει η τριετής διάρκεια. Επίσης, ε, θα πρέπει να προσέξουμε ώστε να μην ε, περιορίσουμε υπερβολικά και με ε, ανόητα προσχήματα τους, τους ε, γεωργούς. γιατί μερικές φορές έχουμε πολύ χαμηλή παραγωγικότητα δυστυχώς. Έχουμε ένα τομέα που πολύ δύσκολα μπορεί να αποθηκεύσει τα προϊόντα του. Γιατί εξαιτία στον αλώσιμο χαρακτήρα Επίση ε, είναι πολύ έθρευστη θέση του απέναντι στου αγοραστέ. Και η εμπορική, στη διαπραγματευτική του ισχύ είναι πολύ σημαντική για να καταλήξουν σε αποδεκτέ τιμέ. Και αυτό η χαμηλή, ο χαμηλό βαθμό οργάνωση του αποδυναμώνει. Θα πρέπει να διασφαλίσουμε αυτή την ισχύ τη συλλογική διαπραγματεύση για του Γιώργους και τι οργανώσει του. Επίσης υπάρχουν κάποιες παράγραφοι που είναι σχετικά σαφείς και φαίνεται ότι αντιβαίνουν στο βασικό κανονισμό. Δεν θα αναπτύξω τώρα διεξοδικά αυτά τα θέματα, θα στείλω γραπτό στις παρατηρήσεις μου στον κύριο Κόρτε και ε, επαναλαμβάνω την προθυμία μου για συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή προκειμένου να προχωρήσουμε και στο κείμενο αυτό. Ευχαριστώ. Ο κύριος Δεκάστρο, παρακαλώ. Ε, Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Οι συνάδελφοι έχουν ήδη εκφράσει πάρα πολλές ανησυχίες που έχει η Επιτροπή μας σε σχέση με τις δύο κατεξουσιοδότηση πράξεις που συζητάμε. Εγώ θα ήθελα να αναφερθώ κυρίως σε αυτά που είπε η συνάδελφος κυρία Ντόρφμαν. Και θα ήθελα να παρακαλέσω τον ε, εκπρόσωπο της Κομισιόν να μας πει το εξής. Ε, σήμερα, κοιτάξτε, ε, ήρθαμε εδώ για να συζητήσουμε γιατί εμείς το ζητήσαμε. Άρα δηλαδή πράγματι το Κοινοβούλιο πρέπει να οργανωθεί καλύτερα. Από την άλλη όμως και το λέω ξεκάθαρα η Κομισιόν είναι εκείνη που θα πρέπει να ενημερώνει καλύτερα την Επιτροπή μας. Γιατί είδατε υπάρχουν ανησυχίες όσον αφορά τα οποροκυπευτικά. Δεν καταλαβαίνουμε γιατί πρέπει να γίνουν κάποιες αλλαγές. Ε, πίσω από τη λέξη απλούστευση ε, κρύβονται κίνδυνοι, ε, μπορεί να υπάρξει αποσύνδεση ε, ή ε, κάποια συγκεντρωμένη προσφορά. αυτη οι κίνδυνοι ε, αναφέρθηκαν στο Τρεντίνο Αλτο Άντιτζε. Εκεί αναφέρθηκε ο συνάδελφος, υπήρξαν προβλήματα, γι' αυτό λοιπόν θα πρέπει να εφαρμόσουμε ακριβώς αυτά που προβλέπει ο κανονισμός για τα απορροκυπευτικά. Αυτή τη στιγμή υπάρχει κίνδυνος να συνδέσουμε να διαλύσουμε τις οργανώσεις παραγωγών, κάτι που το ε, κάναμε, το επιτύχαμε μετά από πολλές προσπάθειες. Όσον αφορά τώρα το κρασί, Κοιτάξτε, θέλουμε να κατανοήσουμε τι ακριβώς σημαίνει αυτή η προσαρμογή στον κανονισμό βάσης. Κατανοούμε ότι είναι απαραίτητο να υπάρξουν παρεμβάσεις στις κατεξουσιοδότηση και τις εφαρμοστικές πράξεις. Εντάξει, σίγουρα εμείς δεν είναι ότι ε, δεν θέλουμε να εφαρμόζουμε τις ε, διατάξεις που προέκυψαν με τη μεταρρύθμιση της ΠΑΚ, αλλά θέλουμε να ξέρουμε και να πούμε ότι δεν πρέπει να καταστρέψουμε αυτά που λειτουργούν καλά και στον ε, στο κρασί από το 2009 και μετά λειτουργούν τα πράγματα σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Τώρα γιατί πρέπει να αλλάξουμε κάτι το οποίο λειτουργεί σωστά. Ε, με χαρά μου ε, θα ακούσω την απάντηση του εκπροσώπου της Κομισιόν. Σας λέω με απόλυτη σαφήνεια ότι αυτοί οι κανονισμοί είναι πάρα πολύ ευαίσθητοι και δεν πρέπει να παίζουμε με τη δυσκολία που έχει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να συμμετέχει στις συνεδριάσεις των εμπειρογνωμόνων. Θέλουμε να ενημερωνόμαστε και όπως μας εγγυάται και η συνθήκη της Λισαβόνας να έχουμε και τη δυνατότητα αρνησικυρίας όσον αφορά αυτές τις πράξεις. Σας ευχαριστώ πολύ. Ε, κυρία Αγγιλέρα. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Ευχαριστώ πολύ για την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για την εξαιρετικά χρήσιμη ενημέρωση. Μιλήσατε για τα όσα έχετε κάνει για τις ε, κατευθυντικές πράξεις που είναι και πολύ σημαντικά. Όπως είπαν και άλλοι συνάδελφοι, θα ήθελα και εγώ να μεταφέρω την ανησυχία μου σε ό,τι αφορά το προσχέδιο με τη μορφή που έχει λάβει σήμερα. Κατά τη γνώμη μου, το σχέδιο πηγαίνει και υπερβαίνει την απλή απλούστευση. Πολλά ζητήματα έχουν αναφερθεί, τα οποία υπερβαίνουν την απλούστευση και που είναι πολύ σημαντικά και απορρέουν από το βασικό κανονισμό. Και περιορίζομαι σε αυτά που αναφέρει το πρώτο σχέδιο. Επιπλέον, η πρόταση αυτή, αν υλοποιηθεί ως έχει, θα δυσκολέψει τις οργανώσεις παραγωγών και δεν θα μπορέσουν να διεκπαιρεώσουν τα επιχειρησιακά προγράμματα. Και οι οργανώσεις παραγωγών, που είναι οι βασικοί συντελεστές, θα δυσκολευτούν για να πραγματοποιήσουν τα επιχειρησιακά προγράμματά τους. Και ο ελάχιστος αριθμός παραγωγών αναοργάνωση θα πληγεί. Επίσης, το θέμα της ε, εμπορίας ε, των τρίτων που δεν είναι μέλη, ε, καθορίζεται ποσοστό για να καθοριστεί να καθοριστούν τα περιβαλλοντικά επιτέγματα των οργανώσεων και επίσης ε, το θέμα της ε, τιμής θέσης στην αγορά. Είναι πολύ σημαντικά αυτά τα σημεία και θα επηρεαστούν από το σχέδιο. Όλες αυτές οι προτάσεις ξεπερνούν κατά πολύ την απλούστευση. Ουσιαστικά τροποποιούν τους κανόνες του παιχνιδιού. Επίσης θίγονται όλες αυτές οι πτυχές, αλλά το πιο σημαντικό αίτημα και της Επιτροπής Γεωργίας και του παραγωγικού τομέα της Ευρωπαϊκής Ένωσης δεν περιλαμβάνεται. Τι συμβαίνει με τις ε, ισχύουσες τιμές απόσυρσης για τις οργανώσεις παραγωγών. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή λέει ότι χρησιμοποιήθηκε μόνο κατά 27% αυτός ο μηχανισμός. Όντω, μπορεί να χρησιμοποιήθηκε λίγο, όχι γιατί οι οργανώσει παραγωγών δεν το ήθελαν, αλλά γιατί οι τιμέ δεν προσαρμόζονται στι ε, παρούσες ανάγκες και στην αξία της ε, τιμής απόσυσης. Γι' αυτό δεν προσέφηκαν στη χρήση αυτού του μηχανισμού. Και ίσως είναι πολιτικό το θέμα, αλλά σίγουρα δεν ε, αναφέρθηκε καθόλου αυτή η πτυχή, παρά τις έντονες επισημάσεις. Και τι θα γίνει με τις τιμές απόσυσης που είναι ένα σημαντικό μηχανισμό για τι οργανώσει παραγωγών. Και γιατί δεν χρησιμοποιείται αυτό ο μηχανισμό, δεν προβληματίζεται η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Επίση, σε ό,τι αφορά την τροποποίηση του καθεστώτο ε, τιμών εισόδου. Γίνονται συνεχείς καταγγελίες για το πρόβλημα με τις ντομάτες από το Μαρόκο. Δεν θα επεκταθώ σε αυτό, το εξήγησαν ε, εμπεριστατωμένα οι προλαλήσαντες. Θα πρέπει να τροποποιηθεί αυτό το σημείο, σίγουρα. Δεν ξέρω ποιο είπε ότι η τροποποίηση δεν έγινε από το Μαρόκο. Είναι μια τροποποίηση που επηρέασε την τιμή του καθεστώτος ε, τιμών εισόδου τη ντομάτα στην Ευρωπαϊκή Ένωση και εξαιτία αυτής της τροποποίηση ε, δόθηκε ευκαιρία στο Μαρόκο να εισάγει ό,τι ποσότητες ντομάτας ε, θέλει, γιατί ε, η τιμή είναι πολύ υψηλή, γιατί ε, βρέθηκε ο μέσο όρο και συνυπολογίστηκε στη τιμή τη ντομάτα και η τιμή τη ντομάτα τσέρι, των μικρών ντομάτων. Εγώ γνωρίζω ότι και στη Μούρσια και στη Γρανάδα οι ντοματοπαραγωγοί απειλούνται με εξαφάνιση εξαιτία αυτή τη κατάσταση που δημιουργήθηκε με το Μαρόκο. Και συμφωνούμε όλοι με την απλούστευση. Όλοι επιθυμούμε την απλούστευση, αλλά οι προτάσεις του σχεδίου σας ξεπερνούν την απλούστευση. Για να μην μιλήσουμε για το ουσιαστικό πρόβλημα που είναι να ενισχύσουμε τους ε, ε, γεωργούς και να ενισχύσουμε τις οργανώσεις παραγωγών. Υπάρχουν κάποιες κανόνες του παιχνιδιού, αυτούς θέλετε φαίνεται να τροποποιήσετε, γιατί αυτό φαίνεται να είναι ο στόχος του σχεδίου. Και διαφωνούμε με αρκετές πτυχές του σχεδίου. Και ελπίζω στι περαιτέρω εργασίε που θα γίνουν και φυσικά και εγώ είμαι πρόθυμη να συνεργαστούμε με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για να βελτιώσουμε το κείμενο προκειμένου να ικανοποιήσουμε τι ανάγκε τη Ευρωπαϊκή Γεωργία. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ κύριε Σαντρία. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Έχουν υποθεί τα ουσιαστικά στοιχεία από τους συναδέλφους μου. Ευχαριστώ και τον κύριο Κόρτε ε, που θέλει να φανεί καθησυχαστικός, παρόλα αυτά βλέπουμε πόσες δυσκολίες υπάρχουν και εντάξει δεν θέλω να τα επαναλάβω γιατί όλα έχουν αναφερθεί. Ιδίως από την κυρία Γιλέρα. Δεν θέλω να επανέλθω στην ντομάτα ή στα απορριπευτικά. Να επισημάνω μόνο κάτι για τον Ίνο. πριν από μερικέ εβδομάδε συναντήθηκα με τον Επίτροπο και νομίζω ότι υπάρχουν πολύ, πολλά προβλήματα και σε άλλους κλάδους σήμερα. Για αυτή την περίοδο τα εξετάζουμε αυτά τα προβλήματα τα οποία δεν πρέπει να τα εξετάζουμε σε κλάδους που ήδη λειτουργούν καλά, όπως είναι αυτός του Ίνου. Και αναφέρατε κι εσείς ότι υπήρξε πολιτική συμφωνία στη μεταρρύθμιση του 2008 και 2013 και πρέπει να μεριμνήσουμε ιδιαίτερως για να μην σπάσει αυτή η συμφωνία. Και να μην χρησιμοποιήσουμε τις εκτελεστικές και καταξιώδεις πράξεις ως πρόσχημα, για να το πούμε έτσι, για να τροποποιήσουμε τελικά από την πίσω πόρτα την υφιστάμενη και κείμενο νομοθεσία. Αυτό θα πρέπει, ε, για αυτό, σε αυτό το σημείο να είμαστε ιδιαίτερα προσεκτικοί και υπεύθυνοι. Και εγώ βεβαίω ε, δηλώνω πρόθυμο να συμμετάσχω στι εργασίε όπω και οι συναδελφοί μου. Γιατί είναι ιδιαίτερω λεπτά αυτά τα ζητήματα. Τώρα, σε ό,τι φορά την επλούστευση, Ναι, θέλουμε να προστατεύσουμε κάποια στοιχεία, αλλά να μην χαλάσουμε και τις ισορροπίες ε, που έχουμε βρει στο παρελθόν, στα παρεγκυφτικά ή στον ίνο. Και ξέρετε ότι και οι επαγγελματίες ε, εξετάζουν ε, με μεγάλη προσοχή τα όσα συμβαίνουν αυτή τη στιγμή. Αυτά ήθελα να πω εν συντομία γιατί πολλά έχουν ήδη υποθεί προηγουμένως. Σας ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Κύριε Κόρτη, σε ευχαριστούμε για την έκθεσή σας. Λέτε ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο δεν συμμετέχει επαρκώς. Εγώ δεν ξέρω γιατί συμβαίνει αυτό. Εγώ ε, μπορώ να μιλήσω μόνο για τον εαυτό μου και να σας πω ότι πολύ ευχαρίστω ε, θα έλεγα τη γνώμη μου γιατί εμείς βρισκόμαστε σε πολύ στενή επαφή με τους αμπελουργούς και τους ε, παραγωγούς απορροκυβευτικών προϊόντων που είναι πολύ σημαντικά στη Γερμανία. Αυτές λοιπόν οι ως είναι πολύ επιφυλακτικέ ως προς τις ε, προτάσεις σας. Ε, το πρόβλημα είναι το ε, έγγραφο εργασίας. Λέτε ότι δεν υπάρχει διαφάνεια, δεν είναι ικανοποιητικό το κείμενο και επίσης λέτε ότι δεν υπάρχουν και συνοδευτικά κείμενα για διάφορες ρυθμίσεις. Κοιτάξτε κύριε Κόρτες, θα χρειαστούμε χρόνο μέχρι να έχουμε όλα τα κείμενα. Για μας όμως είναι καθοριστική σημασία οι αμπελουργοί να μην ε, αντιμετωπίσουν μικρότερη αλλά τουναντίον αντίον ε, μεγαλύτερη ασφάλεια. Αναπέρομαι στον κανονισμό επισήμανσης. Ε, ο κανονισμός αυτός περιλαμβάνει πάρα πολλά στοιχεία από την εμφιάλωση, την επισήμανση και πάρα πολλά άλλα. Δεν πρέπει να βάλουμε εκεί ένα μεγάλο ερωτηματικό. Το έχουμε βάλει και ανησυχούν οι αμπελουργοί. Επίσης ε, αναφερθήκατε και στις ενώσεις παραγωγών οποροκυπευτικών οι οποίοι έχουν κάνει μέχρι τώρα ό,τι ζητάτε σε άλλους τομείς ας πούμε στο γάλα δηλαδή αυτοί ενώθηκαν, έπιαξαν δομές ε, θέσεις εμπορία συνεταιρισμούς, καλές τιμές ε, έχουν καταλάβει καλό μερίδιο στην αγορά τώρα λοιπόν ακούω ότι στο πλαίσιο των δραστηριοτήτων για την προστασία του περιβάλλοντος ε, απαιτούνται περισσότερες ε, ενέργειες από τις οργανώσεις παραγωγών. Και ξέρετε κάτι, αυτό με κατιστά πολύ επιφυλακτική γιατί από ό,τι φαίνεται σε όλους τους τομείς και στον τομέα της ε, προστασίας του περιβάλλοντος αναφέρεστε στα φυτοφάρμακα Τώρα ε, θέλετε να επιβάλλετε και δραστηριότητες προστασίας του περιβάλλοντος. Πώς θα το κάνετε αυτό. Νομίζω ότι πολλοί ε, καλλιεργητές ε, είναι πολύ καλά ενημερωμένοι, συμμετέχουν σε πολλές ε, δραστηριότητες. Το να του ζητάει κανείς και προστασία του περιβάλλοντος, αυτό είναι υπερβολικό. Εγώ πιστεύω ότι πρέπει να βούμε πρακτικά εφαρμόσεις με λύσεις, να προχωρήσουμε, να ενισχύσουμε τους ε, παραγωγούς ε, και να δούμε και λιγάκι κατά πόσο αυτός ο κανονισμός μπορεί να εφαρμοστεί και στην πράξη. Σας ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ κύριο Καπούτο. Sì, grazie. Grazie, Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Θα προσπαθήσω να μην επαναλάβω αυτά τα οποία έχουν ήδη λεχθεί. Ευχαριστώ τον κύριο Κόρτε, τον εκπρόσωπο της ε, Επιτροπής ε, για τις εξηγήσεις που μας ε, έδωσε. Και με αυτή την αφορμή θέλω να καλέσω και τον πρόεδρο να αναπτύξει όλες εκείνες ε, τις ε, δραστηριότητες που πρέπει και που μπορούμε για να επιτύχουμε τελικά μια νέα συμφωνία συνεργασίας. Θέλω λοιπόν να σας πω ότι ανησυχώ πάρα πολύ από όλα αυτά που ελέγχθησαν. Γιατί υπάρχει αυτή η έννοια της ε, απλούστευσης και τελικά πίσω από την απλούστευση κρύβονται όχι απλουστέψεις, αλλά δυσκολίες. Αυτό είναι, ας πούμε, ισχύει για τις ενώσεις παραγωγών. Ε, ας πούμε, υποτίθεται η απλούστευση ε, θέτει ένα αμφιβόλο το θέμα των οργανώσεων παραγωγών, ενώ τα έπρεπε να ε, διασφαλίζει την ε, νομική εξασφάλιση αυτών των ε, οργανώσεων παραγωγών ή έγινε λόγος για προϋποθέσεις που έχουν σχέση με το περιβάλλον προαπαιτούμενα τα οποία προφανώς και πρέπει να διευκρινιστούν αλλά και κατά τη δική μου την άποψη όλα αυτά πρέπει να γίνουν σταδιακά με ένα τέτοιο τρόπο που θα επιτρέψουν την προσαρμογή και τον σεβασμό όλων αυτών των προαπαιτούμενων. Όσον αφορά τώρα τα οποροκυπευτικά, ο Πάολο τα είπε πάρα πολύ ωραία. Γιατί να πρέπει να αλλάξουμε τους κανονισμούς σε ένα τομέα που λίγο πολύ λειτουργεί καλά. Ένας τομέας ο οποίος ε, μεταξύ άλλων ε, έχει δύναμη είναι ισχυρός λόγω του ότι υπάρχει αυτή η διασύνδεση με ε, γεωγραφικές ενδείξεις. Ε, είναι περιττό, ας πούμε, να αποσυνδέσει κανείς ε, τις ε, γεωγραφικές ενδείξεις, τις ετικέτες ονομασίες προέλευσης ε, από τις ε, παραδοσιακές ενδείξεις. Εγώ θεωρώ ότι πρέπει να διατηρηθεί το κείμενο που προβλέπει συγκεκριμένες διευκρινήσεις, όλα αυτά να ισχύουν με ένα και μόνο κανονισμό, γιατί θεωρώ ότι αυτό διευκολύνει τους παραγωγούς. Και δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι όταν θεσπίζουμε κανονισμούς θα πρέπει πάντα να έχουμε κατά νου και εκείνους οι οποίοι δουλεύουν στη γη, στην ουσία δηλαδή. Η κυρία Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Εντάχει να υποβάλω τρεις ερωτήσεις. Η πρώτη αφορά το Μαρόκο. Τι γνώμη έχετε για την απόφαση του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, πώς την ε, λαμβάνετε υπόψη. Επίσης, η απλούστευση στον τομέα των απορροκυπευτικών ε, που είναι το ζητούμενο, πώς θα την υλοποιήσετε και τι μέτρα ρύθμισης θα θεσπίσετε για να αντιμετωπίσετε την κρίση που μαστίζει αυτή τη στιγμή τον κλάδο των απορροκυπευτικών. Και τρίτη ερώτηση για τον Νίνο. Ποιες είναι οι κατευθυντήρες γραμμές που εφαρμόζετε στις εργασίες σας, γιατί από αυτά που άκουσα δεν κατάλαβα να έχετε καμία συγκεκριμένη πρόταση. Δεν έχετε συγκεκριμένη πρόταση για το κρασί. Οπότε ποιες γραμμές σας κατευθύνουν αυτή τη στιγμή για το ίνο, για τον αμπελονικό τομέα. Ευχαριστώ κύριε Σουαζό. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Όταν ακούμε τις επαγγελματίε του κλάδου, η απλούστευση φαίνεται ότι είναι περισσότερο μια πολυπλοκοποίηση περίπλοξη των όνων. Και από το ΚΝΟΚ βλέπουμε ότι και η ε, Εθνική Ένωση Ενοπαραγωγών ε, ΠΟΠ ε, επικρίνουν τα όσα προβλέπονται για την επισήμανση και παρουσίαση των προϊόντων και την πολιτική ποιότητας για τα προϊόντα αυτά. Βλέπουμε λοιπόν ότι δεν είναι πλέον δυνατόν να κάνουμε μια συνολική ανάλυση και για τους ίνους χωρίς ε, γεωγραφική ένδειξη βλέπουμε ότι αναφέρονται και σε μια περιφέρεια πιο μικρή από το κράτος μέλος. Μπορεί δηλαδή ο καθένας να κάνει το οτιδήποτε. Βάσει της Ευρωπαϊκής ε, Ομοσπονδίας ε, των Ίνων ΠΟΠ, τα κρασιά αυτά χωρίς ΠΟΠ θα μπορούν να αποφεληθούν περαιτέρω και έχουμε και αυτό το τομέα της απελευθέρωσης που δεν μα επιτρέπει να αναπτύξουμε τον ανταγωνισμό το οποίο θα πρέπει να γίνει τώρα αναπτύσσοντα και αυξάνοντα τον όγκο. Και όλα αυτά υπό το πρόσχημα της απλούστευσης και έτσι καταστρέφουμε ε, τις ιδιαιτερότητες του νεπραγωγικού κλάδου. Θέλει λοιπόν η Κομισιόν να συνεχίσει την πολιτική της απορρίθμισης σε όλους τους γεωργικούς, γεωργικούς κλάδους παρά και τα κείμενα, παρά και τα συμφέροντα των ε, παραγωγών και των επιλογών των Ευρωπαίων πολιτών και για τους παραγωγούς προεκπαιδευτικών βλέπουμε ότι δεν μπορούμε πλέον να ελέγξουμε τι μπαίνει στην Ευρωπαϊκή Επικράτεια, αλλά για κάποιες ε, χώρες ε, μιλούν και για ε, χώρες μάλλον με πολύ χαμηλό εργατικό κόστος καταφέρνουν να απολούν τα προϊόντα τους σε πολύ χαμηλές τιμές. Και χώρες που δεν είναι μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης όπως η Τουρκία μέσω διάφορων συστημάτων μπορούν να δώσουν πάρα πολλά χρήματα ε, για να ανταγωνιστούν και τα ευρωπαϊκά προϊόντα όπως και στους ε, ανταγωνίζονται σε πολύ μεγάλο βαθμό και τους Γάλλους παραγωγούς που βρίσκονται σε δημοτική κατάσταση. Ευχαριστώ. Κύριε Σέλμπερντες. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Δεν θέλω και εγώ να επαναλάβω αυτά που έχουν ήδη υποθεί. Κύριε Κόρτεπ, Είπατε ότι το Κοινοβούλιο ε, και οι συνεργάτες μας εδώ του Κοινοβουλίου δεν συμμετέχουν στις εργασίες. Κύριε Κόρτε, ε, ξέρετε πολύ καλά ότι εκτιμώ τους εκπροσώπους της ε, Κομισιόν, αλλά κοιτάξτε, όσον αφορά τις συνθήκες της Λισαβόνας, πρέπει να σας πω ότι εκεί έχει γίνει ένα πολύ μεγάλο λάθος. Δηλαδή, μας, μας έδωσαν δικαιώματα το δικαίωμα του να αποφασίζει κυρίω, αλλά δεν μα έδωσαν προσωπικό. Α πούμε, αν δούμε λιγάκι το τι προσωπικό έχουμε εμεί εδώ στην Επιτροπή μα και στα κράτη-μέλη για αυτά τα θέματα που συζητάμε, ε, δεν είμαστε επίση όρει, κύριε Κόρτε. Για πέστε μα λιγάκι εσεί, κύριε Κόρτε, πόσου ε, συνεργάτε έχει η Γενική Διεύθυνση Άγκρη. εμεί έχουμε μια δεκάδα. Και είπα κάποτε στον κύριο Μπαρόζο ότι με βάση τη συνθήκη της Λισαβόνας θα έπρεπε να μας δώσει η Κομισιόν το 5% του προσωπικού της εδώ, να αποσπαστεί αυτό στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για να μπορούμε να εφαρμόσουμε τις συνθήκες της Λισαβόνας. Ίσως πρέπει να το ξανακουβεντιάσουμε αυτό. Κατά τα άλλα, όσον αφορά το θέμα της απλούστευσης, κύριε Κόρτε, εγώ θα σας συνεβούλευα να ε, συμπεριλάβατε τους εμπειρογνώμονες της δικής μας της ε, πολιτικής ομάδας της συζητήσεως και μαζί τους να συζητήσετε τα θέματα των ε, κατεξοδότηση πράξεων. Εμείς ε, ήμασταν οι πρώτοι, οι οποίοι μετά τη συνθήκη της Λισαβόνας ε, θέσαμε έτοιμα για κατεξιδότηση πράξη, ε, συζητήσαμε την Κομισιόν και επιτύχαμε βελτιώσεις στη γεωργική πολιτική. Είναι λοιπόν πολύ σημαντικό το να οργανώσετε κάποια συζήτηση για να καταλήξουμε και σε ικανοποιητικά αποτελέσματα. Επίσης, να επισημάνω και κάτι που το έθιξαν και άλλοι συνάδελφοι. Κοιτάξτε, δεν είναι αλήθεια ότι κάθε απλό απλούστευση, προγραμματιζόμενη επιφέρει και ουσιαστική απλούστευση. Ακούσαμε από την Κομισιόν ότι διάφοροι κανονισμοί για τους σπόρους ε, θα συμπτυχθούν σε ένα κανονισμό. Εμείς όμως απορρίψαμε αυτή την πρόσταυση, γιατί ξέρετε κάτι, αυτή η απλούστευση τελικά θα δημιουργούσε ε, περισσότερες δυσκολίες από ό,τι έχουμε μέχρι τώρα. Όσον αφορά τώρα την κατάσταση στην αγορά, ε, θα ήθελα να παραθέσω κάτι που είπε η κυρία Άστριτ Λούλινγκ ε, πρώην συνάδελφος ε, στην Επίτροπο ε, Μαριάν Φίσερ Μπόλινγκ η οποία είχε πει ότι θα πρέπει κάποιες εκατοντάδες εκτάρια να εξερσωθούν στην Ευρώπη και η κυρία Λούλινγκ ξέρετε τι είχε πει δεν είναι ότι δεν έχουμε αρκετό κρασί στην Ευρώπη μια χαρά κρασί έχουμε μεγάλες ποσότητες μόνο που η κατανάλωση στην περιπολική Ευρωπαίοι πίνουν πάρα πολύ κρασί αυτά είχα να σας πω Πρόεδρος δεν σχολιάζω. No comment. Ο κύριος Φλάναγκαν. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Μία ερώτηση έχω μόνο προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Μήπως θα μπορούσατε να μας εξηγήσετε αυτό που είπατε ε, μικρό ενδιαφέρον η ανάμειξη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Δεν μας ενδιαφέρει απλώς να, να βάζουμε μια σφραγίδα στο τέλος. Μας ενδιαφέρει σε εμπλοκή. Τι ακριβώς εννοούσατε όταν είπατε ότι δεν υπήρχε αρκετή ανάμειξη στο Ευρωπαϊκό Κοινοβουλίο. Ε, θα ήθελα να πω ότι υπάρχει κάτι που πρέπει να το επισημάνουμε. Δηλαδή, με νόμιμα μέσα μπορούμε να καταλήξουμε σε απλούστευση ε, κυρίως όσον αφορά τους ε, παραγωγούς, τους ε, αγρότες. Γνωρίζουμε ότι όσοι έχουν τα πράγματα, κυρίως όσον αφορά το εμπάργο των προϊόντων στη Ρωσία, αυτό θέση ενός πραγωγών είναι καθοριστική σημασίας και όσον αφορά την ονομασία προέλευσης κοιτάξτε ανεξάρτητα ε, με το αν πρόκειται για κρασί ή για άλλα προϊόντα δεν είναι δυνατόν να προβαίνουμε σε εκπτώσεις οφείλουμε να έχουμε πάντα κατά νου τους ε, καταναλωτές οι οποίοι επιθυμούν να γνωρίζουν από πού προέρχονται αυτά τα προϊόντα. Προέρχονται μήπως ε, εκτός, ε, από χώρες εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης ή παρήχθησαν στην Ευρώπη. Στη τελική ανάλυση είναι δικαίωμα του καταναλωτή να γνωρίζει τι προϊόντα καταναλώνει. Sì, grazie, grazie Presidente. Ευχαριστώ πρόεδρε. Να πω μόνο κάτι ε, πολύ μικρό γιατί οι συναδελφοί ε, τα είπαν τα περισσότερα αυτά που μας ανησυχούν. Εμείς σας είπα, ανησυχούμε για το ότι ποτίθεται πίσω από την απλούστευση, κρύβονται άλλοι στόχοι, απορρίθμιση, deregulation σε ένα τομέα ε, σημαντικό ε, στα οποροκυπευτικά δεν ξέρω, ε, τώρα στο κρασί θα μπορούσε να βοηθήσει ε, και στην Ιταλία και τις άλλες χώρες. Ο αγώνας που γίνεται για την υγεία. Ποτίθεται ότι αγωνιζόμαστε για την υγεία, αλλά κατ' ουσίαν θέλουμε να χτυπήσουμε άλλους. Ε, αυτούς που παράγουν κρέας, κρασί, υπάρχουν αυτά. Και Ευχαριστώ τον εκπρόσωπο της Κομισιόν, αλλά θέλω να το ρωτήσω το εξή. Κοιτάξτε, στο έγγραφο εργασία έχουν εξαφανιστεί πάρα πολλές ε, κανονιστικές και ρυθμιστικές ε, αναφορές. Σήμερα μας τα είπατε πολλά προφορικά, αλλά στο έγγραφο εργασία υπάρχει ένα κενό που κατά την άποψή μας ε, αυτό είναι μια πληγή για ένα σύστημα που λειτουργεί καλά. Και ρωτώ το εξή ή λέω το εξή. Η Ευρώπη πρέπει να είναι συνεπή στην αγροτική τη πολιτική. Δεν μπορούμε από τη μια να επενδύουμε στην προστασία των καταναλωτών έτσι ώστε να γνωρίζουν όλοι στην ετικέτα τι περιλαμβάνει το προϊόν και μετά να τους εξαπατούμε για την προέλευση του προϊόντος. Ε, κάποιος όταν αγοράζει ένα προϊόν το συνδέει με μια περιοχή αλλά τελικά μπορεί αυτό να έχει παραχθεί σε τελείως διαφορετικό μέρος. Αυτό είναι πολύ σημαντικό. Το δεύτερο που θέλω να πω είναι το να μην υπάρχει διασύνδεση προϊόντος με συγκεκριμένο τόπο, αυτό είναι πλήγμα ε, για την αγορά. Για τα ελληνικά, ιταλικά, ε, γαλλικά προϊόντα. Οι ε, Γάλλοι το εξήγησαν πολύ καλά, μιλώντας για το terroir, λένε ότι όταν βλέπει κανείς ένα προϊόν, δεν ασχολείται μόνο με, το, με τη χημική του σύνθεση, έχει κατά νου την περιραίουσα ατμόσφαιρα, την ιστορία, ό,τι συνδέει κανείς με αυτό το προϊόν. Εάν λοιπόν αυτά τα εξαφανίσουμε, είναι σαφές ε, ότι αυτό θα ήταν ζημιά. Εμείς ε, ως Ιταλοί το ζούμε αυτό, το ζουν και άλλοι. Θα οδηγούσε σε κακέκτυπα. Αυτό υπάρχει ήδη τώρα. Κακέκτυπα εκτός Ευρώπης. Δεν είναι σωστό θα δώσουμε ένα χειρότερο προϊόν στον καταναλωτή, αλλά και θα επιφέρουμε ένα πλήγμα στην οικονομία που θα είναι πολύ ε, ηχηρό. Σας ευχαριστώ. Ολοκληρώσαμε τον κατάλογο των ομιλητών. Και είναι πολύ σημαντικό ένα τόσο σπουδαίο θέμα ε, που αφορά τα, τις κατεξοδότηση πράξης ε, να το συζητήσουμε εκτενώς. Ήταν πολύ ε, σημαντικό να μην έχουμε περιορισμό στη συζήτηση και να έχουμε εκτενή και διεξοδική συζήτηση. Γιατί πραγματικά το θέμα του κατεξοδότηση πράξεων για τα απορροκυπευτικά και τον ίνο είναι μείζονος σημασία. Ε, και χαίρομαι που είχαμε την πολυτέλεια του χρόνου και δεν χρειάστηκε να το διεκπαιρεώσουμε, να διεκπαιρεώσουμε τη συζήτηση άρων-άρων. Αυτό το θέμα είναι πολύ σημαντικό και αφορά μεγάλο αριθμό παραγωγών στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Γι' αυτό λοιπόν ήταν απαραίτητη τόσο διεξοδική συζήτηση. Θα δώσω τώρα το λόγο στον Διευθυντή Κόρτε για να απαντήσει στις ερωτήσεις των Ευρωβουλευτών επί της ουσίας. Ευχαριστώ και σας ευχαριστώ για τις ερωτήσεις. 16 ευρωβουλευτές ε, έλαβαν το λόγο και θα προσπαθήσω να απαντήσω σε όλα τα επιμέρους σημεία γιατί νομίζω ότι είναι πολύ σημαντικά για το έργο μας. Θα ήθελα, απαντώντας στις αντιδράσεις που άκουσα λέγοντας ότι θα πρέπει να συνεργαστούμε για να βελτιώσουμε το σύστημα και ζήτησα να αναμειχθεί το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο στο έργο και των εμπειρογνωμόνων. Αυτό δεν θα πρέπει να το εκλάβετε ως επίκριση, ως μορφή κατά το προσωπικό της Επιτροπής σας. Το αντίθετο. Έχουμε μιλήσει και διμερώς ε, με πολλούς από εσά και όλοι αναγνωρίζουμε την ανάγκη να βρούμε λύση. Γιατί και εμείς συμφωνούμε ότι θα πρέπει να δίνεται η αίσθηση ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εργάζεται ερήμην του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Επουδενή δεν επιδιώκουμε κάτι τέτοιο. Και το θέμα το κατεξοδότηση πράξεων είναι σχετικά καινούριο είναι εμπειρίες ε, πρωτόγνωρες και συνεχώς ανακαλύπτουμε νέα πράγματα και θέλει και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να συνεργαστεί μαζί σας όσο γίνεται περισσότερο. Αυτό το νόημα είχαν οι παρατηρήσει μου. Σε καμία περίπτωση δεν θα πρέπει να εκλειφθούν ως μορφή για έλλειψη ανάμειξης ή ενδιαφέροντος. Τώρα, προσπάθησα να συνοψίσω τις ερωτήσεις 7-8 σημεία. Οι πιο σημαντικές ερωτήσεις ε, αναφερόταν όπως ήταν αναμενόμενο στον Ίνο, στην επισήμαση του Ίνου και στο έγγραφο εργασία που υπέβαλαν οι υπηρεσίε Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Αυτό το έγγραφο εργασία δεν συνιστά πρόταση. Ήταν ένα copy-paste, μία ε, ε, αντιγραφή και επικόλυση όσων σημείων ε, υπάρχουν στους διάφορους κανονισμούς. Και ήταν λάθος ίσως να το θέσουμε επιτάπητο σε αυτό το έγγραφο εργασία, γιατί πραγματικά δημιούργησε παρεξηγήσει ε, και παρανοήσεις. Και αναλαμβάνω την ευθύνη γι' αυτό. Ήταν ε, λάθος επιλογή να υποβληθεί ε, ως στοιχείο της συζήτησης, γιατί δεν αναφέρεται ο κανονισμός 607 βέβαια στο έγγραφο, δεν γίνεται μνήμα του. Αυτό δεν σημαίνει θέλουμε να τον καταργήσουμε σε καμία περίπτωση. Απλώς Θέλαμε να βολιδοσκοπήσουμε τους ε, εμπειρογνώμονες για να δούμε πώς ε, σε μια προσπάθεια αναδιατύπωση και των 15 κανονισμών. Και κατέστησα σαφές από την ε, πρωινή συζήτηση, αλλά και από άλλες αντιδράσεις, ότι αυτή η μέθοδος δεν λειτουργεί και θα μεταφέρω το μήνυμα στον Επίτροπο, ώστε να αποσύρουμε το κείμενο και να ξαναρχίσουμε από την αρχή ε, δεν βιαζόμαστε και όπως είπαν κάποιοι, αν δεν έχουμε πρόβλημα δεν χρειάζεται να προσπαθούμε να τα επιδιορθώσουμε και όλα. Έχουμε άλλες προτεραιότητες. Το μήνυμα ελήφθη και το κατέγραψα δεόντως. Επουδενή, επαναλαμβάνω, δεν ήταν πρόθεση Ευρωπαϊκής Επιτροπής να ε, αμφισβητήσει προηγούμενες ε, συμβαστικές ε, λύσεις ή πολιτικές συμφωνίες, κύριε Νταντέ, ούτε προς τη μία ούτε προς την άλλη κατεύθυνση. Σε ό,τι αφορά τις τιμές εισόδου και έρχομαι στον τομέα των απορροκυευτικών. Ε, τιμές εισόδου και SIV, δηλαδή Standard Import Values, κατά τιμές αγωγής, κυρίως για τις ντομάτες. Μετά την συμβαστική λύση του 2013 στο βασικό κανονισμό, οι κανόνες άλλαξαν. Οι τελωνιακές διαδικασίες που ίσχυαν πριν το 2013 δεν ισχύουν πια. Οπότε η ε, δεν μπορεί πια να, γίνει, να επαναληφθεί αυτή η υποτιθέμενη απάτη η κατάχρηση εκ μέρου του Μαρόκου. Γιατί δεν ισχύουν πια οι πάλι κανόνε. Σε ό,τι αφορά τι ντομάτε, η κατάσταση στον κλάδο, ιδιαίτερα στην Ισπανία, δεν είναι καθόλου ρόδινη. Για να το πούμε κατεφημισμό. Δεν ξέρω σε ποιο βαθμό αυτό οφείλεται στην αύξηση των εισαγωγών από το Μαρόκο, γιατί έχουμε την αίσθηση ότι η κρίση ε, οφείλεται σε μεγάλο βαθμό και στις προβληματικές καιρικέ συνθήκε που είχαμε στην Ισπανία τον τελευταίο χρόνο. Και αν εξετάσουμε τις στατιστικές των εισαγωγών από το Μαρόκο, βλέπουμε ότι δεν έχουν αυξηθεί τόσο αισθητά. Οπότε δεν είναι αυτές οι αιτίες της κρίσης. Και μάλιστα, ε, όταν ε, υπολογίζουμε τις αποκοπήν μέση εισαγωγή, παίρνουμε το μέσο όρο των ε, βασικών τιμών ντοματών και ντοματινιών. Εκεί δεν έγινε καμία αλλαγή. Το θέμα είναι σκεφτήκαμε αντί να έχουμε ημερήσια καταποκοπή τιμή εισαγωγή, να έχουμε εβδομαδιαία τέτοια καταποκοπή τιμή εισαγωγή, standard import value. Και εξετάσαμε πολύ σοβαρά το θέμα για μακρά περίοδο τις ημερήσεις τέτοιες τιμές SIV και είδαμε τις συνέπειες σε περίπτωση που από την, εβδομαδία, από την ε, ημερήσια περάσαμε σε ένα εβδομαδιαία τιμή. Και είδαμε ότι δεν θα είχαμε διαφορές. Αυτό φυσικά δεν θα ήθελα να γίνει εις βάρος ή με αντίθετη γνώμη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Αν είστε αντίθετοι θα το λάβουμε υπόψη γιατί ακόμη δεν έχει οριστικοποιηθεί καμία απόφαση. Πρόκειται για ένα σενάριο εργασίας ακόμη και όσα σχόλια υποβάλλατε θα τα λάβω πολύ σοβαρά υπόψη. Ό,τι αφορά τις τιμές απόσυρσης ε, στον τομέα των απορροκυπαυτικών στην κατεξοδότηση πράξη δεν προβλέπεται καμία αλλαγή στη συγκεκριμένη κατεξουσιοδότηση πράξη. Γνωρίζουμε ότι οι μέσα απόσυρση είναι ιδιαίτερα χαμηλέ. Ούτε έχουν σκοπό να καλύψουν το κόστο παραγωγή. Και μάλιστα οι τιμέ απόσυρση δεν ορίζονται σε, ε, επίπεδο ώστε να γίνονται, αποτελούν μια εναλλακτική διέξοδο ε, της διανομής, της παραγωγής, αλλά απλώ δίνουν μια ε, δυνατότητα για χρησιμοποίηση του συστήματος και πέραν του γενικού συστήματος απόσυρσης που υπάρχει στο γενικό καθεστώς για τα απορροκυπευτικά υπάρχει και το ειδικό καθεστώς εκτάκτων μέτρων, μέτρων εκτάκτου ανάγκης ε, εξαιτίας του ρωσικού εμπάργου. Και εκεί οι παραγωγοί μπορούν να συμμετέχουν με ευκολότερο τρόπο στο σύστημα απόσυρσης. Υπάρχει και αυτό το καθεστώς, υπάρχει και αυτός ο μηχανισμός, ο ειδικό και θα εξακολουθεί να ισχύει τουλάχιστον μέχρι το φετινό καλοκαίρι. Και στο κείμενο που είδατε δεν υπάρχει καμία αλλαγή στο σύστημα των τιμών απόσυρσης. Τώρα, τα πρόσθετα περιβαλλοντικά κριτήρια και πρόσθετες περιβαλλοντικές απαιτήσεις για τις οργανώσεις παραγωγών στον τομέα των παρακυπευτικών. Ένα σχόλιο που διατυπώθηκε από πολλούς ευρωβουλευτές. Θεωρώ ότι υπάρχει μια παρεξήγηση εδώ, έγινε μια παρανόηση. Ο βασικός κανονισμός, το άρθρο 33 παράγραφος 5 συγκεκριμένα, προβλέπει ότι τουλάχιστον 10% των δαπανών των επιχειρησιακών προγραμμάτων καλύπτουν περιβαλλοντικές δράσεις. Αυτό είναι το νομικό, το νομίμο κριτήριο. Τουλάχιστον 10% των δαπανών των επιχειρησιακών προγραμμάτων καλύπτουν περιβαλλοντικές δράσεις. Αυτό προβλέπει ο κανονισμός. Αυτή είναι η, νόμιμη, νομική υποχρέωση. Το θέμα είναι πώς θα διευκολύνουμε τις ε, οργανώσεις παραγωγών για να εφαρμόσουν αυτό το κριτήριο που υπάρχει, είναι κατοχυρωμένο στο νόμο. Και τι σημαίνει αυτό το 10% γιατί υπάρχουν αφιβολίες. Σημαίνει ότι κάθε κράτος μέλος θα πρέπει... Κάθε μέλο, μάλλον, θα πρέπει να έχει τέτοιο περιβαλλοντικό κριτήριο στι δραστηριότητε. Υπάρχει κάποιο άλλο τρόπο εφαρμογή για τι οργανώσει παραγωγών. Γι' αυτό και προτείνουμε ένα κανόνα που εισάγει μεγαλύτερη ελαστικότητα και λέει τουλάχιστον το 50% των παραγωγών που είναι μέλη της οργάνωσης, τουλάχιστον η μισή δηλαδή θα πρέπει να εφαρμόζουν δύο περιβαλλοντικές δράσεις. Όχι όλα τα μέλη δηλαδή, τουλάχιστον το μισό, το 50% των μέλων. Δεν είμαστε υποχρεωμένοι να το πούμε αυτό στην κατεξοδότηση πράξη, αλλά τι θα συμβεί σε τέτοια περίπτωση κάθε κράτος και κάθε ελεγκτής και κάθε ε, ελεκτική αρχή θα πρέπει να προσδιορίζει τον τρόπο εφαρμογής του κριτηρίου του 10%. Θέλουμε όμως οι κανόνες να είναι οι ίδιοι να ισχύουν ομοιόμορφα σε όλα τα κράτη-μέλη και να μην οδηγούν σε διαφορετικά συμπεράσματα για το πώς εφαρμόζεται αυτό το κριτήριο, αυτή η υποχρέωση του 10%. Και με την πρόταση αυτή προσπαθούμε να διευκολύνουμε τις οργανώσεις των παραγωγών να εκπληρώσουν αυτό το κριτήριο και όχι να τις δυσκολέψουμε. Αν υπάρχουν πάντως άλλες ιδέες να διευκρινίσουμε και να διευκολύνουμε τα πράγματα, πολύ ευχαρίστως να τις εξετάσουμε. Παρόμοιο πρόβλημα έχουμε και με τις οργανώσεις παραγωγών και το θέμα που επισήμαναν πολλοί ευρωβουλευτές, ε, κυρίως από την Ιταλία, για τη δυνατότητα ενός συνεταιρισμού που είναι μέλος μιας οργάνωσης παραγωγών και σε ποιο βαθμό ο συνεταιρισμός μπορεί να θέσει εμπορία τα δικά του προϊόντα εκτός της ε, συντονισμένης ε, ε, στρατηγικής προμήθειας και θέση εμπορίας της οργάνωσης των παραγών. Αυτό το εξετάσαμε διεξοδικά και γνωρίζουμε τη σημασία και τις επιτυχίες που έχουν συγκεκριμένες οργανώσεις παραγών, ιδιαίτερα στην Ιταλία. Και από κοινού με τους εμπειρογνώμονες πιστεύω ότι βρήκαμε μια διέξοδο που θα επιτρέπει σε μια πιο μακροχρόνια περίοδο πριν τη θέση σε ισχύ, όπως είπε ο κύριος Ντόρφαν, να ισχύει. Πάντως κατά τη γνώμη μας δεν έχει αλλάξει ο κανόνας. Ακόμη και σήμερα με τον υπάρχοντα κανονισμό δεν επιτρέπονται τέτοιες πρακτικές. Και σε πολλές χώρες μέλη η αναγνώριση μιας οργάνωσης παραγωγού που έχει ε, ως μέλος ένα συνεταιρισμό που κάνει, έχει τη δική του στρατηγική εμπορία έχει αποσυρθεί φαίνονται περίπλοκα τα πράγματα, αλλά να εξετάσουμε την κατάσταση στα κράτη-μέλη, κάνουμε ό,τι μπορούμε για να εξυπηρετήσουμε καλύτερα τις εργανώσεις των παραγωγών. Δεν χρειάζεται να, πείσετε, να πείσουμε τον Επίτροπο Χόγκαν ή κανένα άλλο υπάλληλο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ότι είναι σημαντικές οι οργανώσεις παραγωγών. Το γνωρίζουμε και μάλιστα τις στηρίζουμε γιατί είναι πολύ σημαντικό να υπάρχουν και είναι ο μόνος μηχανισμό που έχουμε σε έναν τομέα που, όπως είπαμε πολύ χαρακτηρίζεται από μεγάλη αστάθεια και διακύμανση από από αδυναμία αποθήκευση των προϊόντων, οπότε είναι ιδιάζοντα τα χαρακτηριστικά του κλάδου των απορροκυπευτικών και γι' αυτό θα πρέπει να στηρίξουμε τις οργανώσεις των παραγωγών και να τις ε, προαγάγουμε όσο γίνεται περισσότερο. Και μάλιστα δυστυχώ σε πολλές χώρες μέλη είναι χαμηλό ο βαθμός ε, οργάνωσης ε, και συμμετοχής στις οργανώσει παραγωγών. Και είδαμε ότι ήταν πολύ χαμηλός στο σήμερα ο βαθμός οργάνωσης και στο 2004-2007 τα χαμηλότερος. Τώρα αυξήθηκε και εξαιτία του ρωσικού εμπάργου. Θα προσπαθήσουμε να τον ενισχύσουμε ακόμη περισσότερο και κάναμε μια επισκόπηση του γαλακτοκομικού τομέα και εκεί αποφασίσαμε στην αναθεώρηση του πακέτου γαλακτοκομικού τομέα που εμπίπτει στην κοινή οργάνωση αγοράς να υπάρχει δυνατότητα και των παραγωγών των γαλακτοπαραγωγών να ε, συνεργάζονται για κοινή διαχείριση των ε, θεμάτων τους μέχρι 30% ε, της αγοράς. Και ήταν σημαντική αυτή η σύσταση του κυρίου Νταντά για να μας προστατεύσει και να μας θωρακίσει και από τους κανόνες του ανταγωνισμού. Και στην έκθεση που θα υποβάλουμε την Άνοιξη θα δούμε πώς ανταποκρίθηκαν η παραγωγή στην κρίση, στις χαμηλές τιμές και τι μπορούμε να κάνουμε σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Επιτροπής και Ευρωπαϊκής Ένωσης για να βελτιώσουμε την κατάσταση. Και τέλος, ως προς την ερώτηση της κυρία Σένερα για την απόφαση του Γενικού Δικαστηρίου των Ευρωπαϊκών ε, ε, Τη ευρωπαϊκή Ένωση για το μέτωπο Πολυσάριο και την αγροτική, γεωργική συμφωνία με το Μαρόκο. Εμεί αφαισιβάλαμε την απόφαση του πρωτοβάθμιου δικαστηρίου, του Γενικού Δικαστηρίου του Λουξεμβούργου, όπω αποκαλείται. Εφεσιβάλαμε αυτή την απόφαση ε, σε δεύτερο βαθμό κατά της πρωτοβάθμιας απόφαση Αυτά κύριε Πρόεδρε, ελπίζω να τίμησα ε, τους ευρωβουλευτές και να μην αδίκησε κανένα με τις απαντήσεις. Αυτά προς το παρόν. Σας ευχαριστώ. Δεν βλέπω να υπάρχουν συμπληρωματικές ερωτήσεις εκ μέρους των ευρωβουλευτών. Άρα μάλλον καταφέρατε να θίξετε όλα τα ζητήματα που σας επισημάνομαι. Με τη συνθήκη της Λισαβόνας ε, ξεκίνησε μια νέα περίοδος ε, και ε, ισχύουν νέοι κανόνες για τη λειτουργία και εφαρμογή της κοινής γεωργικής πολιτικής. Εξού και η ανάγκη θέσπισης νέων κανόνων και διαδικασιών για την ευθυγράμμιση που απαιτείται. Και πιστεύω ότι είμαστε στο σωστό δρόμο και νομίζω ότι οι ευρωβουλευτές μας ε, είναι και εξοικειωμένοι με το θέμα και καλά ε, ενημερωμένοι γιατί είμαστε εμπειρογνώμονες σε αυτό το τομέα, έχουμε πολύ άμεσες επαφές και με τους γεωργούς μας και νομίζω ότι θα είναι πολύ χρήσιμη και καρποφόρα η συνεργασία με τη Γενική Διεύθυνση Γεωργίας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Ευχαριστώ. Σίγουρα θα επανέλθουμε στα θέματα αυτά γιατί όπως είπαμε είναι πολύ σπουδαία. Και θα ήθελα και πάλι να εκφράσω την ικανοποίησή μου που είχαμε ε, την πολυτέλεια του χρόνου και δεν αναγκάστηκα να περιορίσω το χρόνο ομιλίας των συναδέλφων. Χαίρομαι που στο σημαντικό αυτό θέμα αφιερώσαμε το χρόνο που του άξιζε. Και μία πληροφορία πριν ολοκληρώσουμε, ε, ότι το ΕΛΚ έχει οργανώσει μία συνεδρίαση στη Δευτέρα, 7 Μαρτίου στο Στρασβούργο, 9 ε, με 10 και μισή ε, συνάντηση με τον Επίτροπο Χόγκαν για τη συζήτηση την κρίση, της κρίσης που αντιμετωπίζουν οι γεωργοί. Ε, ένα θέμα που μας επισήμανε ο κ. Νταντά. Ζητήσαμε λοιπόν από τον Επίτροπο να λάβει μέρος σε αυτή την έκτακτη συνεδρίαση της Άγκρη στις 7 Μαρτίου γιατί στις 24 Μαρτίου έχουμε το διαρθρωμένο διάλογο με τον Επίτροπο και πρέπει να γίνει νωρίτερα αυτή η συζήτηση. Και διαλέξαμε την ώρα αυτή 9 με 10 και μισή, ώστε να μπορέσουμε να συμπεριλάβουμε και συζήτηση το θέμα, το θέμα της έκθεσης ε, Ταραμπέλα για την ε, διανομή φρέσκων ε, φρούτων στα σχολεία και μάλιστα πριν την Ολομέλεια και θα συζητήσουμε και το θέμα της ε, υγείας των ζώων. Είναι λίγο αργά 9 η ώρα, 9 με 10 και μισή, αλλά το θέμα είναι σημαντικό. Γι' αυτό παρακαλώ σημειώστε το στα, στις ατζέντες σας ε, για να μην χάσετε αυτή τη σημαντική συνάντηση που θα έχουμε με τον Επίτροπο Χόγκαν. Το απόγευμα έχουμε και την ακρόαση για την αστάθεια των τιμών. Θα διακόψω τώρα τη δημόσια συνεδρίαση της Επιτροπής Γεωργίας. Σας ευχαριστώ για τη συμμετοχή και θα παρακαλούσα τους ε, συντονιστές να παραμείνουν στην αίθουσα, τους συντονιστές ή όλους εκείνους που δικαιούνται να λαμβάνουν μέρος στη συνεδριάση των συντονιστών να παραμείνουν. Οι υπόλοιποι καλό μεσημέρι. Ευχαριστούμε τον εκπρόσωπο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, τον κύριο Κόρτε και Λίωτη δημόσια συνεδρίαση. Περνάμε στη συνεδρίαση των συντονιστών εντός